θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο κύριος Μαριάς είναι ο συντάκτης, είναι ο εισηγητής και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Δράκη. θα σα ήμουν ευγνώμων αν μπορείτε να καθίσετε ή αλλιώ, εάν ησύχως και ηρέμως ε, αποχωρήσετε τις αιθούσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον εισηγητή τον κύριο Νότι Μαριά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το Κοινοβούλιο μας ασκεί μια κορυφαία λειτουργία που προβλέπεται από τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία συνίσταται στην άσκηση δημοκρατικού ελέγχου τη δράση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι ανεξάρτητη ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα δεν σημαίνει και ανεξέλεγκτη ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα. οφείλει λοιπόν η ΕΚΤ να παρέχει λογοδοσία προ το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το μοναδικό ενωσιακό όργανο που εκλέγεται απευθεία από του λαού τη Ένωση, τι προηγούμενε χρονιέ η διαδικασία συζήτηση τη ετήσια έκθεση δράση τη ΕΚΤ στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου περιοριζόταν σε ευχολόγια με απουσία κριτική προ την ηγεσία τη ΕΚΤ και τα πεπραγμένα τη. στην παρούσα έκθεση θέτουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. παρότι έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια από συγκεκριμένε πολιτικέ ομάδε στο πλαίσιο τη επιτροπή οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων με κοινέ συμβιβαστικέ τροπολογίε να αφαιρεθούν σημαντικά σημεία αιχμής που περιείχε η έκθεση που συνέταξα παρότι κάποιοι επιχείρησαν να στρογγυλέψουν τις γωνίες παρότι οι ηρακλείς του στέματος αποδείχθηκαν πιο δραγκιστές από τον κύριο ντράγκη εν τούτης τα κέρια σημεία αιχμής της έκθεσης παραμένουν. η έκτο φίλη να κάνει σημαντικά βήματα προκειμένου να διασφαλίσει ότι κατά την ενάσκηση της αποστολής της δεν θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων λόγω της τετραπλής δράσης που έχει μετατρέψει την έκτη σε κράτος εν κράτη και αυτό γιατί η έκτη υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητος θεσμός άσκησης νομισματικής πολιτικής ενώ ταυτόχρονα υποπτεύει τις 130 μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες της ευρώπης. παράλληλα η έκτη είναι ο μεγαλοδανιστής των χωρών της Ένωση, αφού έχει αγοράσει στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης ομόλογα των κρατών της ευρωζώνης και τέλος είναι μέλος της τρόικας που έχει πτωχεύσει και φτωχοποιήσει τις χώρες του μνημονίου γι' αυτό το λόγο η έκθεση υπενθυμίζει τη σημαντική και συνάμα πρωτοποριακή απόφαση του δικαστηρίου της ευρωπαϊκής ένωσης c 62 δύο που προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφείλει η ect να εκτελεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης μια δικαστική απόφαση που στην ουσία ζητά την έξωση της ect από την τρόικα. ταυτόχρονα η έκθεσή μας ζητά να υπάρξει διαφάνεια και έλεγχος της τρόικας άρα και της ect κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων δίθεν διάσωσης δηλαδή των μνημονίων. κύριε ντράγκη η ανεργία παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ιδίω όσον αφορά του νέου και του μακροχρόνια ανέργου με τα ποσοστά να παρουσιάζουν ιδιαίτερη απόκληση από έξι τέσσερα στη γερμανία σε 26,6% έξι στην ελλάδα και όλα αυτά ενώ η ΕΚΤ και τα κράτη μέλη διέθεσαν αρκετά τρισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης από το δύο και μετά ταυτόχρονα η ΕΚΤ είναι ιδιαίτερα ευμενής στη συνέχιση της άσκησης σκληρής δημοσιονομικής πολιτικής και πολιτικής λιτότητας η οποία μάλιστα δεν μπόρεσε να μειώσει την ανεργία ούτε να μειώσει το δημόσιο χρεο η έκθεση μάλιστα καλεί τα κράτη μέλη να διενεργήσουν λογιστικό έλεγχο του χρέους σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 472 του 2013. Επιπλέον θεωρούμε ότι χρειάζεται μια πολιτική που θα ενισχύσει τις δημόσιες και ιδιωτικέ επενδύσει και θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη αυτό απαιτεί αύξηση ρευστότητας και χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. παρότι η ΕΚΤ ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που ανήλθε στα τέλη του έτους 2015 σε 582 δις ευρώ από τα οποία 17 δις δαπανήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της φτωχοποιημένης Ελλάδος, εντούτοις κύριε Ντράγκη δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς ούτε ο αποπληθωρισμός, ούτε η ανεργία, ούτε η επανάπτυξη. Απέναντι στις αιμονές τη ΕΚΤ για αποδόμηση του κοινωνικού κράτους η έκθεση αναγνωρίζει τα όρια της νομισματικής πολιτικής και επισημαίνει ότι τα οικονομικά προβλήματα της ένωσης μπορούν να αντιμετωπιστούν με δομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες όμως οφείλουν να είναι κοινωνικά ισόρροπες. Από εκεί και πέρα η ποσοτική χαλάρωση και τα χαμηλά επιτόκια δεν μπόρεσαν να συμβάλλουν ούτε στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων ενώ είδαμε ταυτόχρονα να δημιουργούνται προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία που είδαν τις αποδόσεις των αποθεματικών τους να είναι ιδιαίτερα χαμηλές. η έκθεση επικουρεί το πρωταθέν από την κομισιόν πανευρωπαϊκό σχήμα εγγύησης καταθέσεων αλλά επίσης επισημαίνει και τα σημαντικά βήματα που έγιναν για την δημιουργία ενιαίας αρχής εποπτείας των τραπεζών. στο πλαίσιο αυτό επίσης πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η εκτ και για ποιο λόγο επέβαλε πιστωτική ασφυξία στην Ελλάδα από τις αρχές του 2015 και τελικά οδηγήθηκε σε capital controls. Επομένως χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας του ΕΛΑ. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητές για την θετική τους συμβουλή στην έκθεσή μου αυτή. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριο Ντράγκη. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι βουλευτές. Αναμφισβήτητα, σε αυτή τη χρονική στιγμή δοκιμάζεται η συνοχή της Ευρώπης. Καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε ως επιτοπλίστων ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες προκλήσεις. Και γι' αυτό χρειάζεται μια ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση. Με ευγνωμοσύνη επανέρχομαι εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι είναι ένα σύμβολο της ανάγκης που υπάρχει για ευρωπαϊκό διάλογο και ευρωπαϊκές λύσεις. Σήμερα συζητούμε την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2014. Τότε το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μία σειρά από μέτρα για να ανταποκριθεί ε, στην ε, αποδυνάμωση των ε, διάβλων επικοινωνίας νομισματικής πολιτικής και στο περιβάλλον του χαμηλού πληθωρισμού. Οδηγηθήκαμε έτσι σε δύο βασικές μειώσεις σε βασικά επιτόκια εξαγγελίες ε, δράσεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ε, και δύο προγράμματα για ε, στοιχεία ενεργητικού και για καλυμμένα ομόλογα. Το 2014 επίσης άρχισαν οι δραστηριότητες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και άρχισε και ολοκληρώθηκε η συνολική αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Θα ήθελα όμως να στραφώ μάλλον προς το μέλλον στη σημερινή μου ομιλία. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εξηγήσω ποια νομισματική πολιτική εφαρμόζουμε τώρα και γιατί το Μάρτιο θα επανεξετάσουμε τη στάση που τηρούμε. Δεύτερον, θα ήθελα να συζητήσω τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τι χρειάζεται για να τις αντιμετωπίσουμε. Έχω πλήρη επίγνωση των σημαντικότερων ζητημάτων για αυτούς που καταρτίζουν την πολιτική αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η οικονομική επιτυχία φυσικά είναι μέρος της λύσης σε άλλους τομείς. Και γι' αυτό η άμβλυνση των οικονομικών κινδύνων οφείλει να είναι ύψιστη προτεραιότητα για τους πολιτικούς ηθήνοντες. Πριν από τρία χρόνια περίπου άρχισε να αποκλίνει ο πληθωρισμός από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ γύρω στο 2%. Από τον Οκτώβριο του 2013 είναι κάτω του 1% ο πληθωρισμός. Κατά το 2015 ο βασικός πληθωρισμός, χωρίς τα τρόφιμα δηλαδή και τα ενεργειακά προϊόντα, στην Ευρωζώνη ήταν πολύ χαμηλός ή και αρνητικός ε, λόγω των χαμηλών προϊόντων βασικών αγαθών και έτσι εκτιμήθηκε στο 0,4% τον Ιανουάριο του 2014 στην Ευρωζώνη, ο ετήσιος πληθωρισμός βάσει του δίκτυου τιμών καταναλωτή. Εκ παραλλήλου, έπρεπε διαρκώς να αναθεωρούμε τις προοπτικές για τον πληθωρισμό. Ενώ στις αρχές του 2015 γινόντουσαν προβλέψεις για τον πληθωρισμό μέχρι 1,5% το 2016 και 1,8% το 2017, το Δεκέμβρη προέβλεψαν ένα επιτόκιο μόνο 1% για το 2015 και 1,6% για το 2017. Με αυτά τα δεδομένα αποφάσισε το Δεκέμβρη η ΕΚΤ να δράσει και πάλι. Δύο άξονες έχει η αποτίμηση της νομισματικής πολιτικής από πλευράς μας. Πρώτον, παρατηρούμε ότι τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί από το καλοκαίρι του 2014 ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Η νομισματική τόνωση της οικονομίας μέσα από αυτά τα μέτρα οδήγησε σε ευρία χαλάρωση των συνθήκων χρηματοδότησης, τονώθηκε η παροχή πίστης και έκτοτε έχει χορηγηθεί ουσιαστική στήριξη με στόχο την ανάκτηση ανάκαμψη της Ευρωζώνης. Απουσία αυτών των μέτρων η Ευρωζώνη θα έχει οδηγηθεί σε καθαρό αποπληθωρισμό πέρυσι και θα είχαν ακόμη ταχύτερα ε, κατακριμνιστεί οι τιμές ε, και η ανάπτυξη θα ήταν σαφώς ε, χαμηλότερη. Δεύτερον, κρίνουμε αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα. Όντως, όμως ταυτόχρονα είναι και ανεπαρκή σε σχέση με τις επιδεινούμενες πρακτικές σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών. Υπήρχε ένας συγκεκριμένος κίνδυνος, δηλαδή χωρίς να αυξήσουμε την τόνωση με την ποσοτική χαλάρωση, ε, ο πληθωρισμός δεν θα ε, πανερχόταν στο μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% ε, μέσοπρόθεσμα. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να προσαρμόσουμε την νομισματική μας πολιτική. Μειώσαμε και πάλι το επιτόκιο αποδοχής από πλευράς της ΕΚΤΕ στο μείον 0,3% και η καταληκτική προθεσμία για τις αγορές ε, κάθε μήνα προβλέπεται για το τέλη Μαρτίου 2017 ενώ διατηρείται η αιρεσιμότητα για τις προοπτικές ως προς τον πληθωρισμό και επίσης θα επανεπενδύσουμε τις βασικές πληρωμές από τα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού μόλις οριμάσουν για όσο χρειαστεί. Επίσης θα συνεχίσουμε τις βασικές ε, δράσεις αναχρηματοδότησης ε, και τις ε, τριμηνιές δράσεις αναχρηματοδότησης σε σταθερά επιτόκια βάσει διαγωνισμών για όσο χρειαστεί και τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τελευταίας περίοδου διατήρηση των αποθεματικών το 2017. Από τότε που συνεδριάσαμε στις αρχές Δεκεμβρίου άλλαξαν και πάλι τα δεδομένα μέτρια η ανάκαμψη στην ε, Ευρωζώνη και στηρίζεται βασικά στην εγχώρια ζήτηση. Όμως έχουν ε, αυξηθεί οι κίνδυνοι για ε, ύφεση της οικονομίας και πάλι υπάρχει μεγαλύτερη ανασφάλεια σε σχέση με τις αναπτυξιακές προοπτικές των αναδυόμενων οικονομιών ε, και υπάρχει μεγάλη πτυτικότητα στις αγορές ε, χρηματοπιστωτικών ε, αγαθών και αγαθών και επίσης γεωπολιτικοί κίνδυνοι προστίθενται σε αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι η το έσχατο κύμα αποπληθωρισμού βασίζεται στην νέα μεγάλη μείωση των τιμών πετρελαίου ταυτόχρονα υπάρχουν χαμηλότερες προβλέψεις σε σχέση με τον πληθωρισμό και γι' αυτό θα πρέπει να επανεξετάσουμε τους διάβλους που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε ε, να επηρεάσουμε μελλοντικά τις τιμές και τη μισθολογική πολιτική τελικά στις οικονομίες της Ευρωζώνης. Και γι' αυτό στην τελευταία μας συνεδρία στον Ιανουάριο κρίναμε ότι ε, Συντρέχει ανάγκη αναθεώρησης, ε, ε, επανεξέταση και επαναπροσδιορισμού ενδεχομένως τη νομισματική μας πολιτική, ε, στις αρχές Μαρτίου όταν οι νέε μακροοικονομικέ προβλέψει θα είναι στη διάθεσή μας. Η νομισματική μας πολιτική λειτουργεί αισίω και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συμβάλλει αυτό που της αναλογεί ούτως ώστε η ανάκαμψη να συνεχίσει. Όμως ελοχεύει ο κίνδυνος και αν τελικά επαληθευτεί αυτό θα μπορούσαν οι συνθήκες να υπονομεύσουν αυτή την πολιτική μας. Είναι μεγάλες προκλήσει που αντιμετωπίζουμε και σχετίζονται με την ε, παγκόσμια κατάσταση, την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οικονομικές, δημοσιονομικέ πολιτικέ των κρατών μελών και η πολιτική αστάθεια σε σχέση με το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρώτον, σε σχέση με τι παγκόσμιε συνθήκε. Ε, οι αναπτυξιακέ προοπτικέ, ε, αργά αλλά σταθερά βελτιώνονται σε ανεπτυγμένε οικονομίε. Το αντίθετο συμβαίνει όμω σε αναδυόμενε οικονομίε. Επίση, η ανάπτυξη είναι σε ιστορικά χαμηλά, οι αναδυόμενε αγορέ αντιμετωπίζουν οικονομικού και χρηματοπιστωτικού κινδύνου ε, λόγω διαρθρωτικών και μακροοικονομικών προβλημάτων και ανισορροπιών ε, και έτσι χρειάζεται να προσαρμοστούν και μειώνουν τι τιμέ των βασικών αγαθών. Είναι ευπαθεί λοιπόν αυτές οι οικονομίες και ε, δεν μπορούν να προσαρμοστούν παρά μόνο με αυστηρότερες ε, χρηματοπιστωτικές πολιτικές. Ε, βασικό ζήτημα είναι ποιε θα είναι οι επιπτώσεις για αυτές τις αναδυόμενες οικονομίες με αυτές τις αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης και με τις μειωμένες εκροές κεφαλαίου και σε ποιο, σε ποιο βαθμό αυτό θα επηρεάσει επίσης την τις αλλαδαπές επενδύσεις ε, για τις ε, οικονομίες της Ευρωζώνης. Θα χρειάζεται ανθεκτικότητα λοιπόν για την ε, οικονομία της Ευρωζώνης. Δεύτερον, χρειαζόμαστε απαντήσεις ως προς την πολιτική σε σχέση με τα, τις χρηματοπιστωτικές μας αγορές. Ε, υπήρχαν διάφορα επεισόδια κόπωσης στο δεύτερο ήμιση του 2015 και αυτό δείχνει ότι έχουμε επιτύχει πολλά με την Τραπεζική Ένωση, όμως δεν έχει αυτό, αυτή η προσπάθεια προσπάθεια ολοκληρωθεί. Για να είναι υγιές το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα πρέπει να σημειωθεί η πρόοδος σε δύο αλληλένδετους ομολογουμένους τομείς. Πρώτον, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και να εφαρμόσουμε τα όσα ξεκινήσαμε με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και τον ενιαίο μηχανισμό εκαθάρισης τραπεζών, διότι αυτή είναι η βασική πυλώνες Τραπεζικής Ένωσης. Έτσι χρειαζόμαστε περαιτέρω νομοθετικές ε, κανονιστικές διατάξεις για την εποπτική αυτή δράση, εξασφαλίζοντας έτσι και μια ε, συνεπή εφαρμογή της οδηγίας BRRD για την ανάκαμψη και την εκαθάριση των ε, τραπεζών. Επίσης χρειαζόμαστε ένα βασικό απόθωμα για το ενιαίο Ταμείο Εκαθάρισης για να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία του και επίσης θα πρέπει να υπάρχει εξίσου υψηλή εμπιστοσύνη όλα τα κράτη-μέλη για τις καταθέσεις. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Μείωση λοιπόν των κινδύνων, επιμερισμός των κινδύνων είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και θα πρέπει να επιδιώκουμε παράλληλα αυτούς τους δύο στόχους. Είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. Τρίτον, Υπάρχουν οι προκλήσει που σχετίζονται με τι δημοσιονομικέ και οικονομικέ πολιτικέ ε, των κρατών μελών που χρειάζονται αποφασιστική δράση ω προ την πολιτική. Έτσι θα συμβάλλουμε στην οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συμμορφωθούμε πλήρω με τι απαιτήσει ε, του Συμφώνου σταθερότητα και Ανάπτυξη. Αυτό είναι σημαντικό για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη που υπάρχει στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και την αηφορία των δημοσιοοικονομικών. Επίση, ε, οι χώρε θα μπορούσαν να υποφεληθούν από μια ε, φιλοαναπτυξιακή σύνθεση και μίξε των δημοσιονομικών πολιτικών. Έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ως προς τα δημόσια οικονομικά και το φορολογικό σύστημα θα είναι φιλικότερο ως προς την ανάπτυξη. Με την κυκλική ανάπτυξη της Ευρωζώνης ε, θα πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας με αποτελεσματικές διεθνωτικές πολιτικές για να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον παρέχοντας ε, τις απαιτούμενες δημόσιες υποδομές. τέτοιου δράσεις είναι ζωτική σημασία για να αυξήσουμε ε, τις παραγωγική, επενδύσει, παραγωγικές επενδύσεις, να τονώσουμε δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Εάν ε, με προσοχή και σωστό σχεδιασμό εφαρμόσουμε τις σωστές μεταρρυθμίσεις, τα θετικά αποτελέσματα ταχύτατα θα τα διαπιστώσουμε, κυρίως ως προς την υποστηρικτική στάση μας σε σχέση με την νομισματική πολιτική. Τέταρτον και θα κλείσω, υπάρχει πολιτική πολιτική αστάθεια σε σχέση με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αυτό ισχύει στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία λύση που θα γύρωνε και πάλι το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επέτρεπε ε, στην, ε, την περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωζώνης ε, θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση επίσης είναι μια αρχιτεκτονική που παραμένει δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι πολίτε και οι αγορές δεν έχουν την ασφάλεια που απαιτείται σε σχέση με την ικανότητα που έχουμε να αναλάβουμε από κοινού τις ευθύνες μας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να τι αποδείξουμε το αντίθετο. Κλείνοντας ε, θα ήθελα να επανέλθω στο υποσυζήτηση θέμα, ε, δηλαδή το ψήφισμα για την ετήσια έκθεση για το 2014. Σας διαβεβαιώ ότι αποδίδουμε την δέουσα σημασία σε αυτό το έγγραφο, μα θυμίζει, θυμίζει το καθήκον μας να με διαφανή τρόπο, με λογοδοσία να επιτελούμε τα καθήκοντά μας. Η δημοσίευση των πρακτικών των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου που αρχίζει αυτό το μήνα είναι ένα μόνο από το παράδειγμα αυτής της δεσμευσής μας. Προσβλέπω στη σημερινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντράγη. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον αντιπρόεδρο της, κυρία, της Επιτροπής, τον κ. Ντομπρόφσκης, ο οποίος θα λάβει αμέσως τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κρητικής Τράπεζας, έντιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Μαριά <clears throat> και τους συναδέλφους του στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση αυτή αυτή η ex ε, έκθεση για την δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σημαντικό στοιχείο δημοκρατικής λογοδοσίας και συμπλήρωμα των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Ευρωπαϊκή Κομισιόν συμμέριστε την άποψη του Κοινοβουλίου για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως αναφέρεται στις συνθήκες και είναι απαραίτητο να συνεχίσει να ασκεί το ρόλο της για την επίτευξη της ε, σταθερότητας των τιμών. Η νομισματική πολιτική είναι στην αποκλειστική τη αρμοδιότητα με τις ε, ενέργειες των τελευταίων ετών, όπως είναι η μειώση των επιτοκίων και οι μακροχρόνιες ενέργειες αναχρηματοδότησης και επίσης και η αγορά στοιχείων του ενεργητικού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αντιμετωπίσει τον στόχο της να έχει πληθωρισμό σε, στα πλαίσια των στόχων της. Όλα αυτά λοιπόν έχουν εξασφαλίσει την αποτροπή της, του χρηματοπιστωτικού κατακαιρματισμού. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να διατηρήσει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%, κάτω από το 2% αλλά κοντά στο 2%. Η προσπάθειά της για την οικονομική ανάπτυξη ε, αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ε, εξελίξεις όπως είναι η μείωση της τιμής του πετρελαίου και η μείωση της οτιμίας του ευρώ που είναι ιδιαίτερα θετική για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς. Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή κλειδονισμούς ιδίως από την ανατολική γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γεωπολιτικό επίπεδο και έχουμε και την επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μειώσουν τις προβλέψεις για οικονομική μεγέντηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχουμε τροποποίηση τις οικονομικές μας προβλέψεις για το ε, επόμενο έτος. Η Κομισιόν συμμερίζεται απόλυτα της απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βασίζεται μονάχα σε, στην νομισματική πολιτική και ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να αυξηθεί η οικονομική μεγέθυνση και να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας. Θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες διαφορετικές αλλαγές και να εφαρμοστούν αυτά κάτι μέλη. Οι διαφορετικές αλλαγές στην νομισματική και δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να γίνουν για να εξασφαλιστεί μια καλύτερη προσαρμογή στην ζήτηση και, και μέτρα για την τόνωση της προσφοράς, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μειώσουν τα ελλείμματά τους και να σταθεροποιήσουν το επίπεδο χρέους τους. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν ακόμα μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις που, ζητούν, που απαιτούν δημοσιονομικές προσαρμογές από αυτές. Η Κομισιόν συμφωνεί λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η δημοσιονομική προσαρμογή με την χρήση της ευελιξίας που βρίσκονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να συνοδευτούν και από μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, στις αγορές εργασίας, ώστε να αναζωογονηθεί η ανταγωνιστικότητα, να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί το κλίμα του επιχειρήν. Η Κομισιό λοιπόν θεωρεί ότι αυτό είναι και μια προτεραιότητα και συγκεκριμένα το το σχέδιο επενδύσεων, το EFCI, θα μπορέσει να βοηθήσει ιδιαίτερα την ανάκαμψη και να, να εξασφαλίσει καλύτερη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Κομισιό λοιπόν έχει υποστηρίξει αυτό το σχέδιο και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητε προπαρασκευαστικέ ενέργειε για την λήψη αποφάσεων για τα θέματα αυτά στην Ευρώπη. Με όλα τα, τα διοικητικά εργαλεία και κυβερνητικά εργαλεία του Ταμείου αυτού να είναι στη θέση τους, είναι έτοιμο να λειτουργήσει αυτό το ταμείο και έχουμε κάθε διαβεβαίωση ότι ο στόχος των επενδύσεων 315 δισεκατομμύριων ευρώ θα επιτευχθεί μέσα στην τριετή περίοδο που προβλέπεται. Η Κομισιόν επίσης συμμερίζεται την άποψη του Κοινοβουλίου για την Ένωση Κεφαλαιογορών. Θέλουμε να ενισχύσουμε την πολυμορφία των πηγών χρηματοδότησης, να ευνοήσουμε την δυνατότητα χρηματοδότησης από την κεφαλαία αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδίω. Είναι ένα φιλόδοξο στόχο λοιπόν η Ένωση Κεφαλαιογορών και η Κομισιόν βασίζεται στην υποστήριξη και τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι αντίστοιχε νομοθετικέ διαδικασίε. Συγχρόνω, συμφωνούμε με το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να παραμείνουμε επάγρυπνοι για του κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα που παρουσιάζονται στι τωρινέ συνδικέ τη αγορά. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να κλείσω υπογραμμίζοντας το ότι βλέπω πολύ κοινό έδαφος μεταξύ των δικών σας απόψεων και της Κομισιόν. Με καθησυχάζει το ότι μπορούμε εμείς να βασιζόμαστε στην υποστήριξή σας στον αγώνα μας για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω σε μια πλήρη και οικονομική συζήτηση σήμερα. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης. Καλησπέρα σας, συνάδελφοι, χαιρετώ και τον ε, κύριο Ντράγκη. Ξεκινούμε με τις δηλώσεις των πολιτικών ομάδων. Ο λόγος τον κύριο Φάντα Κέλαρε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγκη, η σύνταξη αυτής της έκθεσης δεν ήταν κάτι το απλό. Οι συζητήσεις ήταν θερμές. Μιλούσαμε για πολλά διαφορετικά ζητήματα και για τις διαστάσεις που έχει πάρει το χρήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ευτυχώς αυτά δεν έφτασαν ως την σύνταξη της έκθεσης. Θα έπρεπε οι εθνικοί υπουργοί λοιπόν να πάρουν αποστάσεις και να μην παρεμβαίνουν στη δική σας χάραξη πολιτικής. Η γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παραμένει καθοριστική για την ευρωπαϊκή οικονομία και θα πρέπει να μην επηρεάζονται οι ε, διευθυντές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι διοικητές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα εθνικά κράτη. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να παραμείνουμε έντιμοι στη συζήτησή μας, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο δεν ε, θέλουμε να, να έχουμε εδώ κάποια κορόιδα που μπορεί να είναι μικροκαταθέτες ενώ τα, οι μεγάλοι καρχαρίες θα εποφελούνται ανενόχλητοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να ισχύει και για τους μικρούς καταθέτες και για τους ε, μεγάλους ε, επιχειρηματίες πρέπει να, αυτούς που μπορεί να είναι δανειστές, πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι του παιχνιδιού. Κάποιοι επίσης θα ήθελαν δράνεια. Είναι πολύ πιο εύκολο αυτό από το να αναλάβουμε δράση. Χρειάζεται μια ισόρροπη δράση και το ίδιο και π.χ. η σύνταξη της έκθεσης. Ευχαριστούμε. Από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κ. Μαυρίδης. Κώστα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά να συγχαρούμε τον εισηγητή τη έκθεση παρά τι όποιε διαφορέ τον κύριο Μαριά. Κύριε Ντράγκη, καλωσορίσατε. Ε, η παρουσία σα στην Ολομέλεια είναι πάντα ευπρόσδεκτη γιατί ενισχύει μεταξύ άλλων και τη δημοκρατική νομιμότητα. Καταρχά αναγνωρίζουμε τι προσπάθειε που καταβάλλετε και επικροτούμε την πολιτική σα ειδικά με το πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση, σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα ε, και περιβάλλον για τον πληθωρισμό και επιστροφή στην ανάπτυξη. Εν τούτης, η Ευρωζώνη είναι ακόμα μια έθραυστη και ένα ανιομογενές πεδίο με πολιτικές και κοινωνικές αποκλίσεις. Γι' αυτό και καλωσορίζουμε πρόσφατα την δήλωση του κυρίου Κερέ, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές αποκλίσεις στην Ευρωζώνη και μίλησε για τα κράτη εκείνα τα οποία θα έχουν πλεόνασμα και θα πρέπει να προβούν σε περισσότερες δημόσιες επενδύσεις. γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα τη δική σας δήλωση σε αυτό το θέμα. Ε, δεύτερον ο χρηματοπιστωτικός κατακαιρματισμό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στην ευρωζώνη. Το κόστος, δανεισμού για τις μικρές και μισέ επιχειρήσεις παραμένει ψηλότερο από τις μεγάλες, ιδίως σε εκείνα τα κράτη-μέλη που είναι σε οικονομική κρίση και τα πράγματα γίνονται διπλά δύσκολα. και εδώ θα ήθελα τη δική σας άποψη για τον τρόπο παροχής χαμηλού κόστους προς την πραγματική οικονομία. ένα άλλο θέμα τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο λόγω και των ιδιαίτερων αρχών λειτουργίας τους και την αποστολή τους. θα πρέπει οι εποπτικές αρχές να έχουν υπόψη τους ότι υπάρχουν ειδικέ αρχές που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και θα ήθελαμε και το δικό σας σχόλιο. τέλος με δύο σύντομα σχόλια. πρώτον μη εξυπηρετούμενα δάνεια. ποια είναι η δική σας θέση θα πρέπει να υπάρξει ένας κατάλληλος μηχανισμός όπως στην ισπανία και ιρλανδία ή κάτι άλλο. και μια τελευταία κουβέντα για τις καταθέσει και την προστασία τι προτίθεστε να κάνετε για εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία δεν θα ακολουθήσουν τις δικές σας υποδείξεις και θα έχουν την Τραπεζική Ένωση ΑΛΑΚΑΡΤ. Σα Σας ευχαριστώ. Από του συντελετικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Όζοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σεκητά, συνάδελφοι, κύριε Ντράγκη, η έκθεση εξετάζει τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για την οποία ακούστηκαν πολλέ επικριτικές φωνές. Χρειαζόμαστε εργαλεία που να λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα ώστε να τονωθεί η οικονομία της Ευρώπης και προφανώς πρέπει να αναζωογονήσουμε την πραγματική οικονομία και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η ΕΚΤ αναλαμβάνει τέτοιες δραστηριότητε και θέλει να παραμείνουν οι μακροοικονομικέ συνθήκε αλλά και οι ιδιωτικέ και δημόσιε επενδύσει σταθερέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει όλοι αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν. Τότε θα ήταν καλύτερο το οικονομικό περιβάλλον και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενθαρρύνουμε ταυτόχρονα και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όσον αφορά την έκθεση για τι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου είναι το εξή ο ανεξάρτητος χαρακτήρας της λήψης αποφάσεων στην ΕΚΤ και ο ρόλος εποπτείας που έχει αναλάβει, ιδίως ό,τι αφορά την νομισματική πολιτική. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων της ΕΚΤ. Ευχαριστούμε από τους φιλελεύθερους η κυρία Φαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα θερμό καλωσόρισμα προς τον πρόεδρο Ντράγκη και τον ε, αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Μαριά και τους σκιώδεις εισηγητές. Σας ευχαριστώ για την πολύ αρμονική συνεργασία που είχαμε για την έκθεση αυτή. Ε, στην έκθεση αυτή το Κοινοβούλιο εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την ποσοτική χαλάρωση. Ε, τα 60 δις που φαίνεται να είναι σαν αυξητική ορμόνη για την ε, ανάπτυξη η οποία θα σώσει το σώμα της οικονομίας. Κύριε Ντράγκη, δεν αρκεί όμω η νομισματική πολιτική αυτή καθεαυτή. Χρειάζονται και οικονομικέ μεταρρυθμίσει, όπω καταλαβαίνουμε. Και το αναφέρετε και στο τρίτο σημείο τη παρουσίασή σα ε, σήμερα το απόγευμα, ότι κάτι πρέπει να γίνει ε, στι οικονομίε μα. Συμφωνείτε λοιπόν μαζί μου ότι δεν πάνε όλα ε, τα οικονομικά στοιχεία προ τη σωστή κατεύθυνση. Σε κάποιε χώρε οι αγορέ εργασία φαίνεται να έχουν παραλύσει και μοιάζει να μην έχει γίνει καθόλου η μετάβαση από το δουλεύω για να ζήσω στο δουλεύω για να έχω μια ζωή ε, ρυθμισμένη. Έχουμε λοιπόν ε, μεγάλα ελλείμματα και πολλές εντάσεις με μικρή, αύξηση, με μικρή ανάπτυξη της οικονομίας και υψηλή ανεργία. Πολλές χώρες δυσκολεύονται για να τα βγάλουν πέρα. Οπότε προκύπτει το εξής ερώτημα μπορούμε να συνεχίσουμε και να τονώνουμε, να επενδύουμε στην προσωπική χαλάρωση, υπάρχουν παράπλευρες συνέπειες. Και για τα συντεξιωτικά ταμεία και για την οικονομία γενικώ και επίσης οι τιμές του πετρελαίου. Χωρίς αυτές δεν είναι τόσο δραματικά χαμηλός ο πληθωρισμός. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε σε αυτόν τον βαθμό ποσοτικής χαλάρωσης. Σίγουρα χρειάζονται γεωργικέ μεταρρυθμίσει και συγκεκριμένε οικονομικέ πολιτικέ, στοχευμένε. Όμω δεν δέχονται πιέσει αυτή τη στιγμή έτσι όπω έχουν διαμορφωθεί. Αρκεί μόνο ποσοτική χαλάρωση. Ευχαριστούμε για την κούβα, κύριο Ντεμάζη, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριο Δράγκη είπε whatever it takes, θα κάνω ό,τι χρειάζεται και έχει καταπραγίνει τι ε, χρηματαγορέ. Αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για τις Ιταλικές ε, τράπεζες και η κρίση στην ευρωπαϊκή αγορά συνεχίζεται. Έχουμε λοιπόν ένα λόγο για όλα αυτά. Είχατε πει στο Jackson Hall κύριε Δράκη ότι υπάρχει έλλειψη δημοσίων ε, επενδύσεων για να ενισχυθεί η νομισματική πολιτική. Οι τράπεζες με τη μείωση των δανείων δεν δίνουν δεν δίνουν καθόλου δάνεια και χρηματοδότηση και επενδύσεις παρά το γεγονός ότι είναι μηδενικά τα επιτόκια αυτή τη στιγμή δεν φτάνει το χρήμα αυτό στην αγορά, αλλά δημιουργεί περαιτέρω φούσκες. Λέμε ότι θα πρέπει να είναι 2% ο πληθωρισμό, αλλά οι Financial Times κορόιδεψαν του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτε λέγοντα ότι ο στόχο πρέπει να είναι περισσότερο κοντά στο 0,1-0,2. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει σε δυσκολία το ευρωπαϊκό νόμισμα και είχε πει στους επενδυτές στην Ιρλανδία, στι τράπεζε στην Ιρλανδία ότι έπρεπε να ακολουθήσουν τα μέτρα τη γιατί αλλιώ θα βγουν έξω από το ευρώ. Και το ίδιο έγινε στην Κύπρο. Τελικά καταλήγουμε στο να καταλαβαίνουμε ότι είναι η λιτότητα ανόητη, ότι αυτό είναι το πραγματικό σύνδεμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αγοράσει τα ομόλογα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλιώ κινδυνεύει να κατακαιρματιστεί η Ευρώπη και να χαθεί το ευρώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ λεπτό, συνάδελφοι, να τελειώσουμε με τις επίσημες δηλώσεις των πολιτικών ομάδων και μετά έχουμε τρόπο να ακουστούν και όσοι έχουν ζητήσει γαλάζια κάρτα. Κύριος Ουρτάσουν για 1,5 λεπτό για την ομάδα των Πρασίνων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δράγη, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αυτό το κοινοβούλιο σας έχει καλωσορίσει και εσά και τα μέτρα που έχετε λάβει πάρα πολλέ φορές ε, στα μέτρα μη συμβατικής νομισματική πολιτική έχει χαιρετήσει τη θέλησή σας να συνεχίσετε την αγορά στη δευτερευγενή αγορά κρατικών ε, ομολόγων. Παρ' όλα αυτά πολλές φορές τα προγράμματα αυτά κύριε Ντράγκη και το πρόγραμμα της ε, ποσοτική χαλάρωσης ήρθαν κατόπιν εορτή και όχι με τον τρόπο με τον οποίο θέλαμε. Παρά τον τεράστιο όγκο του δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο επίπεδο τιμών, όπω είπαν οι συναδελφοί μα και στον πληθωρισμό. Και επίση το πρόγραμμα αυτό δεν είναι στοχευμένο ώστε να μπορέσει να φτάσει πράγματι στην πραγματική οικονομία, όπω έχουμε ζητήσει πάρα πολλέ φορέ. Περισσότερο δημιουργεί φυσαλίδε φούσκε κερδοσκοπικέ και δεν ενισχύει την πραγματική οικονομία. Ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά μόνο με την νομισματική ε, πολιτική. Δεν υπάρχει πολιτική η οποία να μπορέσει να υποστηρίξει τη συνολική ζήτηση σε δημοσιονομικό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν. Για να κλείσω κύριε Δράγη, τη στιγμή που εμεί αξιολογούμε το αργό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να μιλήσουμε και για την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σαφέ νομικό πλαίσιο για την ΕΛΑ, για την, για την έκτακτη αρρωγή ε, Αυτό γίνεται με τρόπο αυθαίρετο. Εξαρτάται από την πολιτική ε, κατεύθυνση μια κυβέρνησης και μόνο. Και στην περίπτωση της ε, Κύπρου πάλι ελήφθησαν αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παράλληλα με αυτά τα οποία γίνονται στο Eurogroup. Όλα αυτά έθεσαν σε μεγάλο κίνδυνο την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε ο κύριος Βάλη για την ομάδα της Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι δράσεις της ε, ΕΚΤ για το 2015 είναι ένα προσχεδιασμένο ε, πρόγραμμα από πολύ καιρό. 330 εκατομμύρια άτομα έχουν, ε, πολίτες δηλαδή, έχουν παραδώσει την νομισματική τους κυριαρχία στην ΕΚΤ και το τραπεζικό σύστημα το ίδιο. Οι λαοί έχουν πλέον ε, χάσει τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και βρίσκονται υπό τη δικτατορία των Βρυξελών και της Φραγκφούρτης. Η ΕΚΤ δημιουργεί το πρώτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης, τον δημιούργησε μέχρι το 2014 για να εξυπηρετήσει συμφέροντα και αποτυχημένες νομισματικές πολιτικές των επιμέρους τραπεζών, αλλά και το ίδιο με την εποπτεία των ε, κεντρικών τραπεζών. Επίση, ε, δηλώνει και χαράζει νομισματικέ πολιτικέ και οικονομικέ πολιτικέ που δεν τι ε, ανήκουν, όπω με τα δημοσιονομικά των κρατών, τι προλογικέ πολιτικέ ή τι επενδύσει. Όλα αυτά οδηγούν σε διασπάθηση δημόσιων πόρων και οδηγούν σε ιδιωτικοποιήσει. Το 2016 θα έχουμε ύφεση παγκοσμίω με την αύξηση των μεταναστών και την οικονομική επιβράδυνση παγκοσμίω. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούν αυτές οι προσωπικότητες που δεν έχουν εκλεγεί άμεσα να εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαών, όπως ε, θα έπρεπε να σημειώνει και η έκθεση των αντιπροέδρων. Είναι ένας ακόμη κόλαφος ε, στο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε μια νέα δημοκρατική μορφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση με δημοκρατικές κινήσεις έστω και συντονισμένες από το ευρώ. Δεν είναι το ενιαίο νόμισμα και η έκτο στόχος στόχο τη Ευρωπαϊκή και αυτοί που την επερασπίζονται με θρησκευτική ευλάβεια την οδηγούν σε αποτυχία. Ευχαριστούμε η κυρία Άνεμαν για 1,5 λεπτά για την ομάδα των Εθνών και τη Δημοκρατία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, μετά από 7 χρόνια κρίση στην ευρωπαϊκή οικονομία, είδαμε ότι οι φιλελεύθεροι και οι χριστιανοδημοκράτε. έχουν επηρεάσει μέχρι και τη σύνταξη της έκθεσης του κυρίου Μαριά για να δώσουν ένα σύγχρονο χάρτη στον κύριο Ντράγκη. Ε, εδώ ε, ακόμη και αν ήταν πολύ επιφυλακτικός ο κύριος ε, Ντράγκη, ο κύριος Τούσκ είπε ότι η ΕΚΤ αγόρασε εθνικά ομόλογα ξεπέρασε την εντολή της. Εδώ έχουμε φτάσει να είμαστε ευνοχισμένοι και το δόγμα ντράγκη όλα πάνε καλά να καθαγιάζει το ευρώ. Αυτά που έχουν συμβεί όμως είναι πραγματικά χειρότερα. Θα πρέπει να δούμε αν ο κύριος Ντράγκη μπορεί να εξακολουθήσει την πολιτική του χρέους, της ανεργίας και της ε, μετασφοράς ε, των ε, χρημάτων των καταθατών στα χέρια των διοικητών. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν τονώνει την ανάπτυξη ούτε βελτιώνει τις συνθήκες ζωής. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι από αυτά τα θέματα εξαρτάται η επιβίωση των συμπολιτών μας, από την επιβίωση την ίδια του ευρώ. Η πολιτική σας έχει προκαλέσει το χάος και μας οδηγεί στην άβυσο και στην ε, κατάρρευση την οικονομική. Γιατί να πρέπει να σωθεί αυτό το νόμισμα. Ίσως αν σταματούσατε εδώ κύριε Ντράγκη να ήταν πιο ευφυές και πιο σκόπιμο. Με συγχωρείτε, κύριε Άνεμανς, δεν μπορείτε να προσβάλλετε δημοσίως τους ε, υπόλοιπους, κυρίως τους προσκεκλημένους μας. Ο κύριος Συναδεινός για ένα λεπτό από τους μη ανεγραμμένους. Κύριε Πρόεδρε, μία και μόνο φράση της έκθεσης απεικονίζει την ουσία της ύπαρξης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και την οικονομική πολιτική της Γερμανίας και κατ' επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράγραφος 11 επικροτεί την κατηγορηματική δέσμευση τη ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του ευρώ την οποία ανέλαβε τον αύγουστο του. δύο τα πάντα για το χρήμα όχι για του πολίτε ούτε τα έθνη ούτε καν για τι χώρε. η ελλάδα πέρσι διαπραγματεύονταν με του θεσμού για την επιβίωσή τη. η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα πιστή στην πολιτική τη ανεξαρτησία σταμάτησε την παροχή ρευστότητα προ τη χώρα μου για να επιβάλει την εκδικητική συμπεριφορά των ευρωπαίων στον κακό μικρό υποτιθέμενο αδερφό του. είναι φανερό ότι η λεγόμενη σταθερότητα του ευρώ είναι απλά ένα μέσο επιβολής των οικονομικών συμφερόντων της γερμανίας άρα μέρος του προβλήματος. για να γίνει μέρος της λύσης πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση η ευρωπαϊκή ένωση και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με εθνικιστικές κυβερνήσεις που ενεργοποιούν τον πολίτη την οικογένεια και το έθνος έναντι στο χρήμα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ομάδων, τώρα θα περάσουμε στις γαλάζιες κάρτες. Μία αναπληκτή. Κυρίως ε, Ροζάτη για μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ κατά τη γνώμη μου επικεντρώθηκε σωστά στην αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών και στην συμβολή προς την σταδιακή ανάκαμψη ε, της Ευρωζώνης. Εμείς συμβατικά μέτρα όπως ε, τα αρνητικά επιτόκια ε, και η αγορά στοιχείων ενεργητικών έπρεπε να έχουν ε, αναλυθεί ως μέτρα νωρίτερα και θα είχαμε τότε καλύτερα αποτελέσματα. Ε, όμως δεν απευθύνω καμία κριτική κύριε Τράκη διότι γνωρίζω ότι έχετε πολιτικούς περιορισμούς και συναντάτε ισχυρότατη αντίσταση από κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι τα, δεδομε γεγονότα τα ίδια σας επαλήθευσαν ε, την ε, ορθότητα των ε, μέτρων αυτών και διέψευσαν τους αντιπάλους σας. Είναι ισορροπή η έκθεση που συζητούμε σήμερα. Είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το πρώτο σχέδιο που συζητήσαμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και κατά τη γνώμη μου ήταν γεμάτη από αδικαιολόγητες επικρίσεις κατά της έκτια θέματα για τα οποία δεν είναι αρμόδια θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ε, σε μία από τις προηγούμενες συναντήσεις ε, στα πλαίσια του νομισματικού διαλόγου με την ΕΚΤΕ είπατε θα εξετάσετε το ενδεχόμενο του ελικοπτέρου, δηλαδή η παροχή μετρητών στους παίκτες ε, της αγοράς. Τι πιστεύετε γι' αυτό ως προς την νομική βάση για τις θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου αν υιοθετηθεί. Κύριε Ροζάτη, υπάρχει γαλάζια κάρτα για σας. Τη δέχεστε, κύριε Βαντάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ροζάτη, ωραία τα είπατε τώρα. Είπατε για τον κύριο Τράγη ότι επιτέλεσε πολύ καλά το καθήκον του. Μα με ξαφνιάζεται. Δεν καταλαβαίνω. Ο στόχος είναι η σταθερότητα των τιμών και ο πληθωρισμός πρέπει να είναι στο 2%. Εδώ και χρόνια όμως δεν έχουμε επιτύχει αυτό το επίπεδο. Πώς ακριβώς έκανε σωστά τη δουλειά του ο κύριος Τράγκη. Δεν το καταλαβαίνω. Ροζάτη, έκανε ό,τι ήταν δυνατό και ό,τι ενέπτε στην ε, εντολή του βάσει των συνθήκων. Είπα όμως ότι θα μπορούσαν αυτά τα μέτρα να έχουν αναλυθεί νωρίτερα και είπα ταυτόχρονα ότι υπήρχαν οι περιορισμοί ε, πολιτικής φύσεως, αλλά ο τελικός απολογισμός, διότι μας δείχνει ότι με τα μέτρα του Μάριο Ντράκη, όπως είπε το 2012, will do whatever it takes, θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να επανέλθει στην ανάπτυξη Ευρωζώνη. Αυτό το πέτυχε. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Γκουαλτιέρη τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες για τη συνεισφορά του για να βελτιωθεί η έκθεση αυτή, ένα κείμενο ισόρροπο, όπου με σαφήνεια εκφράζεται μια θετική αποτίμηση για την πολιτική και οικονομική νομισματική δράση της ΕΚΤ αναγνωρίζεται η σημασία των μη συμβατικών μέτρων που ε, προωθήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Σημερίζομαι και την αξιολόγηση του Πρόεδρου Ντάγκη για τις ε, μακροπρόθεσμες εξέλιξεις στο μακροοικονομικό σκηνικό Θέλουμε ενίσχυση της εσωτερικής οικονομίας, κυρίως ε, ε, βάσει της κατανάλωσης, ενώ βλέπουμε γύρω μας μια αποδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομίας με μια επιβράδυνση στις αναδυόμενες οικονομίες, κάτι που προκαλεί βεβαιότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Βέβαια δεν μπορούμε να επιδράσουμε εύκολα στην παγκόσμια αγορά, μπορούμε όμως να κάνουμε πράγματα για την Ευρωζώνη. Καταρχάς προχωρώντας και προσαρμόζοντας τα μέτρα της νομισματικής πολιτικής και ε, αυτό είναι πολύ θετικό καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ομόφωνα δήλωσε έτοιμο να συνεχίσει την προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση για να επιτευχθούν οι προαναγγελθέντες στόχοι. Η νομισματική πολιτική δεδαμόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την μετάβαση από μια κυκλική εξέλιξη σε μια διαρθρωτική ανάπτυξη. Χρειάζονται και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με κοινωνική ισορροπία προκειμένου να ε, τονωθεί το δυναμικό αύξησης και ανάπτυξης της οικονομίας μας. Ταυτόχρονα πολιτικές των συναθρισμένων προπολογισμών πρέπει να συμβαδίσουν με την νομοσματική πολιτική και όχι να αντίκυνται σε αυτήν. Όσοι έχουν φορολογικέ δυνατότητε πρέπει να τι αξιοποιήσουν και όσοι έχουν λιγότερο περιθώριο θα πρέπει να ακολουθήσουν με έναν ρυθμό βιώσιμο, εφαρμόζοντα όλου του κανόνε του Συμφώνου Σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένη τη ευελιξία που, που αυτό εμπεριέχει. Επίση, πρέπει να συμπληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση έτσι περαιτέρω, έχοντα μια μακροπρόθεσμη θεώρηση ε, τη ε, έκθεση των πέντε προέδρων του Fiscal Backstop και επεξεργαζόμενη την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εγγύηση των καταθέσεων. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα επηρεάσουν και το διεθνέ πλαίσιο, έχοντα υπόψη και τι ανάγκε τη οικονομική σταθερότητα. Ευχαριστούμε κύριε Γκουαλτιέρη, κύριο Λούνα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δράγη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πράγματι είναι ανεξάρτητη, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να λογοδοτείτε για την πολιτική σα. Στο τέλο του προηγούμενου χρόνου, ο επικεφαλής οικονομολόγος σας απήντησε σε 7 ερωτήματα που του θέσανε και η απάντησή του ήταν ότι θα δοθεί 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για την αγορά στοιχείων ενεργητικών. Αλλά δεν ανέβηκε παρόλα αυτά ο πληθωρισμός <clears throat> ελέγχθη ότι θα υπάρξει ποσοτική χαλάρωση χωρίς περιορισμούς. Αλλά με τον τρόπο αυτό δημιουργείται φυσαλίδες, φούσκες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χωρίς να βοηθάτε την πραγματική οικονομία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω αυτά που είπε ο William White, ο οποίος είπε ότι η νομισματική πολιτική είναι πολύ λιγότερο λειτουργική σε τέτοιες περιπτώσεις και οι αντικές επιπτώσεις αντίθετα είναι πιο μακροπρόθεσμες. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να σκεφτούμε αυτά που είπε ο αναλυτής αυτός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλβέτ ε, Τσαμπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θέλω ευχαριστώ τον κύριο Δράγη και τον κύριο Επίτροπο. Τέσσερις ιδέε βασικές σε ένα λεπτό. Θα ήθελα να σας πω κύριε Δράγη ως τεχνικός των τραπεζικών θεμάτων ήσασταν πολύ καλός. Αλλά ένα άλλο ερώτημα. Δεν σας ε, ανησυχεί το ότι όλα αυτά τα οποία έχει κάνει η Κίνα έχουν γίνει σε βάρος του ευρώ στα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα η είσοδο τη Κίνα, παραδείγματο σε βάθο του ευρώ. Δεύτερον, εμεί υποστηρίζουμε πάντα το γεγονό ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα ούτε την παραγωγικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε πάρα πολλέ μεταρρυθμίσει οι οποίε είναι εκκρεμεί και πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Επίση, ω τεχνικοπολιτικό ε, τραπεζικό, θέλω να σα ε, εξάρω το έργο σας για τα πρώτα βήματα που κάνετε για την εγγύηση των καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι πάρα πολύ άτολμα και πάρα πολύ βραδεία, βραδέα αυτά τα βήματα. Επίσης, ως ε, Ευρωπαίος Τραπεζίτης το 2014 εξασφαλίσετε να υπάρχουν τεράστια κέρδη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Καλό είναι αυτό αλλά γιατί <clears throat> δεν σκέφτεστε περισσότερο για το πώς αυτά τα κέρδη της ΕΚΤ μπορούν να βοηθήσουν να υπάρξει καλύτερη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαδημούλης για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη και κύριε Ντομπρόφσκης, δεν αρκεί η νομισματική πολιτική. Χρειάζεται και αλλαγή οικονομικής πολιτικής. Και γι' αυτά πρέπει να απαντήσει και ο παρόν κύριος Ντομπρόφσκης. Γιατί απαιτείται εγκατάλειψη της μονομερούς λιτότητας και στροφή στην ανάπτυξη. Τόνωση των επενδύσεων και της ζήτησης, ιδιαίτερα στις πλεονασματικές χώρες κύριε Ντομπρόφσκης, γιατί καθυστερεί η πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων που είναι ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου της τραπεζικής ενοποίησης, ως πότε θα βάζει βέτο ο κύριος Σόιμπλε. Κύριε Ντράγκη, σκοπεύετε να προχωρήσετε και να ενισχύσετε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ή θα το μαζέψετε επειδή έχετε εσωτερική αντιπολίτευση από υπερσυντηρητικούς κύκλους που εκφράζει ο κύριος Βάιτμαν. Και πότε επιτέλους θα μετάσχει και η χώρα μου η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και πότε θα πάψει να δανείζεται με μεγαλύτερα επιτόκια από ό,τι άλλες χώρες. Υπάρχουν ενδείξεις σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει και εσείς να πάρετε πρωτοβουλίες για να μην στραγγαλίζετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδημούλη. Υπάρχει ερώτηση για σας με γαλάζια κάρτη, κάρτα από τον κύριο Σοφοζέρ. Την δέχεστε παρακαλώ κύριε Σοφοζέρ. Oui, cher collègue. Pourquoi... Ναι, αγαπητέ συνάδελφε, γιατί δεν ζητάει η ελληνική κυβέρνηση να κόψει νόμισμα η ΕΚΤ για να επενδύσει στις ε, Ανανεώσουμε πηγές ενέργειας, να επενδύσει στην ελληνική οικονομία, γιατί τότε θα επενδύαμε στην πραγματική οικονομία, αντί να φτιάχνουμε πλάστα, ε, πλαστό νόμισμα. Γιατί ποσοτική χαλάρωση δεν περιορίζεται μόνο στις τράπεζες. Ευχαριστούμε κύριο Παπαδημούλης για την απάντηση. Η διάλυση της ζώνης του ευρώ και η επιστροφή στα εθνικά νομίσματα είναι το πρόγραμμα της Μαρή Λεπέν όχι της κυβέρνησης Τσίπρα. Η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ ήταν το σχέδιο του κυρίου Σόιμπλε, που ευτυχώς ακυρώθηκε το καλοκαίρι. Η ελληνική οικονομία σταθεροποιείται και εκτιμούμε ότι το επόμενο διάστημα και από το δεύτερο εξάμεινο του 2016 θα περάσουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό που χρειάζεται και γι' αυτό αγωνιζόμαστε εμείς από την αριστερά είναι όχι η διάλυση της Ευρώπης αλλά η αλλαγή της Ευρώπης, η κοινωνική Ευρώπη. Ο κύριος Φλίν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Ντράγκη, λέτε ότι οι πολιτικές σας αποδίδουν. Όμως, οι κακές επιδόσεις στην Ευρωζώνη είναι στο φως των προβολέων, διότι ε, αυτή τη στιγμή δεν είναι μάλλον στο φως των προβολέων, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε την καταστροφή του χώρου Σέγγεν και όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα καταραίει. Ε, αυτά που συμβαίνουν με το Σέγγεν ε, μας φέρνουν ε, φρικιαστικότερες εικόνες ε, στους τηλεοπτικούς δέκτες, αλλά οι συνέπειες και δική σα πολιτική είναι πολύ σαφή, όπως ε, το 40% ενεργεία στην Νότια Ευρώπη και η καταστροφή του εργασιακού δυναμικού με διαρκή επιβράνηση της, νοσοκο... οικονομίας. Η ποσοτική χαλάρωση μπορεί να χρειάζεται για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα στο Νότο, όμως αν εφαρμοζόταν σωστά θα ήταν και πάλι ένα πολύ μικρό βήμα για να διορθωθούν οι ανισορροπίες που υπάρχουν λόγω των διαφορών στην οικονομική ισχύ των ε, επιμέρους κρατών. Το κάθε κράτο χρειάζεται το δικό του νόμισμα για να μπορεί να καθορίσει τα επιτόκια του, το ε, ισοζύγιο, το εμπορικό ισοζύγιο, όπως κάθε χώρα πρέπει να μπορεί να ελέγξει τα σύνορά τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μονό για ένα, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να καταγγείλω κυρίως την στάση των μεγάλων πολιτικών ομάδων και την πίεση του στον εισηγητή τον κύριο Μαριά που ουσιαστικά αλλίωσαν την, το περιεχόμενο της έκθεσής του. Μία λέξη η οποία δεν έχει αναφερθεί είναι το θέμα του, της τιμής του πετρελαίου. Πριν από 1,5 χρόνο ήταν σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και με τον τρόπο αυτό υπήρξε μία αποσταθεροποίηση της, ε, του πετρελαιακού τομέα και της τραπεζικής, του τραπεζικού κλάδου. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή με την πτώση της τιμής του πετρελαίου ένα μεγάλο κίνδυνο από η μείωση των τιμών κατά 50% λοιπόν μέσα σε μερικές εβδομάδες δεν έχει να κάνει με την, ε, με την ε, προσφορά και τη ζήτηση στι αγορές πετρελαίων αλλά έχει να κάνει μονάχα με την κερδοσκοπία στα παράγωγα πετρελαίου. Έχουν <clears throat> λοιπόν για κάθε συναλλαγή που γίνεται στην πραγματική αγορά αλλάζει χέρι το ίδιο βαρέλ πετρελαίου 200 φορές κάθε μέρα στο, στην αγορά παραγωγών. Θα πρέπει να σταματήσει λοιπόν αυτή η τεράστια διακύμαση που οφείλεται στην κερδοσκοπία. Όλα αυτά περιπλέκουν περισσότερο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την επίτευξη του στόχου του 2% <clears throat> για, την, ε, για τον πληθωρισμό. Και αυτό θέτει σε κίνδυνο και την φερεγγιότητα των μεγαλοσυστημικών τραπεζών. Η κερδοσκοπία στα παράγωγα για τα βασικά προϊόντα και η αντιμετώπιση της ήταν από τα κύρια από τους κύριους στόχους της ε, γαλλικής κυβέρνησης που ήθελε να ηθικοποιήσει τον καπιταλισμό. Αλλά αυτό δεν έγινε. Κύριε Δράγκη, λοιπόν, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την κερδοσκοπία στις τιμές της ενέργειας και να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών ενέργειας στη ζώνη του ευρώ. Ευχαριστώ. Στο Λογιάν. <coughs> για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι χωρίς τις αποφάσεις οι οποίες ήταν επαγγελματικές και στεναρές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ευρωπαϊκή οικονομία, η οικονομία της ζώνης του ευρώ, θα είχε παραμείνει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα στην ε, στασιμότητα και στον αποπληθωρισμό. <clears throat> Αλλά δεν έχουμε σταθεί αρκετά στο αντίκτυπο της πολιτικής του φτηνού ευρώ για τις μακροχρόνιες ε, επενδύσεις και για τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν συνολικά στο θέμα των αποταμιεύσεων. Τα συνταξιδοτικά ταμεία, οι ασφαλιστικοί φορείς, οι επενδύτες θεσμικού χαρακτήρα, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μακροχρόνιες επενδύσεις θα χάσουν λόγω αυτής της πολιτικής. Και πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα που πολλοί ήδη θέτουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για πόσο χρονικό διάστημα θεωρείτε ότι η νομισματική σας πολιτική, η οποία οδηγεί σε χαμηλό ευρώ, μπορεί να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φερέιρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Επίτροπε Ντομπρόσκη, Πρόεδρε Ντράγκη, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, ε, κύριε Ντράκη, που μου στείλατε, διότι ε, ε, είχα συντάξει την έκθεση για τη διαδικασία με τους πέντε προέδρους και περιμένω ακόμη τις απαντήσεις των υπολείπων προέδρων. Πήρα απάντηση μόνο από εσά. Θα ήθελα να τονίσω ε, πόσο σημαντικός είναι ο μηχανισμός διάσωσης ε, των ε, τραπεζών και σήμερα υπενθυμίσατε ότι είσαστε πεπισμένος πως αποθεματικό για το Ταμείο Εκαθάρισης και Σταθεροποίηση των Καταθέσεων είναι ζωτικά στοιχεία της πολιτικής σας. Ελπίζω όμως και η Επιτροπή και το Συμβούλιο να τηρήσουν τις δικές τους δεσμεύσεις σε αυτό το τομέα. Έχουμε ενιαίο υποπτικό μηχανισμό από τον Εύριο του 2014 και έχουμε και ενιαίο μηχανισμό εκαθάρισης και όλα αυτά τα στοιχεία σταθεροποίησης ε, της Τραπεζικής ε, Ένωσης ε, δεν επαρκούν διότι έχουμε τον, το σύστημα εκαθάρισης το οποίο στην πράξη δεν έχει εφαρμόστεί και με την οδηγία BRDD διαπιστώνουμε πάρα πολλά προβλήματα κυρίως στην περίπτωση ευπαθών οικονομιών. Σε μια τέτοια οικονομία όταν χρειάζεται ενίσχυση ενίσχυση των κεφαλαίων για τις ιδιωτικές τράπεζες βλέπουμε ότι ε, για πρώτη φορά δεν επαρκούν τα μέτρα γιατί υπάρχουν απώλειες για τους καταθέτες σε άλλες διαδικασίες εκαθάρισης. Δηλαδή ε, στέλνουμε ε, αντικρουόμενα μηνύματα στις αγορές ενώ θέλουμε να μεταβούμε στην Τραπεζική Ένωση και διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση είναι επισφαλέστερη σε σχέση με το παρελθόν. Κυρίως για τις ευπαθείς οικονομίας διότι υπάρχουν σοβαρότατοι συστημική κίνδυνη και έτσι τίθενται πάρα πολλά ερωτηματικά. Ποια είναι τα βασικά, ποιος παρακολουθεί αυτές τις επιπτώσεις των μέτρων, τις παρακολουθεί η ΕΚΤΕ ή το Συμβουλίο Συστημικού Κινδύνου ε, στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ε, τι γίνεται, υπάρχει ε, για τα κόκκινα δάνεια συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση τους. Ναι, ολοκληρώνω. Και τελικά υπάρχει συνολικό όραμα για το τραπεζικό σύστημα των κρατών μελών, ε, διότι έχουμε αφήσει την πολιτική ανταγωνισμού στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τελικά αναλαμβάνει τα ενία ή έκτε με τον ενίο εποπτικό μηχανισμό. Α δοθούν κάποιε απαντήσει ε, γιατί μπορεί να είναι μοιραίε οι εξελίξει για την Ευρωζώνη αν δεν λειτουργήσουν τα μέτρα τη έκτε. Σα ευχαριστούμε. Η κυρία Φωνστόρ, ένα λεπτό. Ja, heute reden wir μιλάμε σήμερα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις πρωτοβουλίες της, την παρουσία του κυρίου Ντράγκη. Εσείς εδώ και πολύ καιρό ακολουθείτε μια πολιτική εθνικών συμφερόντων. Σώζουμε χώρες που είναι αφαιρέγγες και τράπεζες οι οποίες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν. Αλλά αυτό είναι δημοσιονομική πολιτική, δεν είναι νομισματική πολιτική, δεν έχετε καμία εντολή να το κάνετε. Το 25 Σεπτεμβρίου 2012 είπα θα κάνετε ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί το ευρώ. Μα δεν είναι δικιά σας υπόθεση αυτό κύριε Ντράγκη. Εσείς πρέπει να κρατήσετε την αξία του ευρώ σταθερή και όχι τον αριθμό των κρατών μελών που είναι στην Ευρωζώνη. Και τώρα λέτε ότι θα συνεχίσετε τις προσπάθειές σας και θέλετε να στοχεύσετε καλύτερα στον, στον πληθωρισμό. Κάποιος θα πληρώσει τώρα όμως αυτήν την πολιτική σας. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν την κρίση, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ασφάλειες ζωής και άλλου είδους επενδύσεις και αποταμιεύσεις. Οι απλοί άνθρωποι αυτοί θα πληρώσουν την ύφη. Η πολιτική σας δεν λύνει το πρόβλημα και πλήττει τους απλούς ανθρώπους. Αυτό είναι άδικο και, δεν είναι, και, είναι και αντικοινωνικό και δεν είναι μια καλή υπηρεσία για την Ευρώπη. Ο κύριος Φλάνεγκαν, για ένα λεπτό. Κύριε Ντράγκη, ε, έκθεση για τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ιρλανδία μετά από τις σχετικές ανακρίσεις δακτυλοδεικτούν την ΕΚΤ με νέα δίψη που θα μπορούσαν να έχουν διασωθεί με τα ομόλογα τα οποία δεν ήταν εγγυημένα και αυτό λόγω των δραστηριοτήτων του προκατόχου σας, του κυρίου Τρισέ. Εννέα δις που χάθηκαν λοιπόν, πέταξαν, μεγάλη αδικία για την Ιρλανδία που αυτή τη στιγμή ε, είναι κάτω από την επίβλεψη του ευρώ και το αναφέρει και η Eurowatch. Ε, αυτά τα ομόλογα, ε, κύριε Ντράγκη, ε, ουσιαστικά ξοδεύτηκαν για να σώσουν μόνο τους μετόχους κάποιων τραπεζών και να προστατεύσουν το ευρώ για τράπεζες που δεν ήταν συστημικές. Οι τράπεζες αυτές τελικά ε, καθαρίστηκαν όμως αυτά τα 31 δις ε, από την κεντρική μας τράπεζα πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία. Έξι λοιπόν δις που θα αναγκαστεί να δανειστεί η τράπεζά μας, συν άλλα 25 που θα είναι το νέο δάνειο. Απαντήστε σε αυτή την ερώτηση, σας ρωτώ απευθεία σήμερα. Μπορείτε να συνεργαστείτε συνεργαστείτε μαζί μα για να σταματήσει αυτή η χιδεότητα. Μην επιτρέψετε να διαπραχθεί αυτή η αδικία για την Ιρλανδία και για τα παιδιά μα. Απαντήστε σε αυτή την ερώτηση για μια πρώτη φορά σε αυτό το κοινοβούλιο. Μια έντιμη ερώτηση να απαντηθεί. Η κυρία Κάπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, Πρόεδρε όταν έχουμε μια αποδυναμωμένη ε, ανάπτυξη στην Κίνα, αυτό οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη διακύμανση σε ε, παγκόσμιο επίπεδο. Αν δούμε λοιπόν και ποιο είναι το αποτέλεσμα το, της ποσοτικής χαλάρωσης και της αγοράς αξιογράφων, αυτά δεν έχουν οδηγήσει σε μια ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι, εξακολουθεί να είναι χαμηλός ο πληθωρισμός, πολύ μακριά από το 2%, πολύ κοντά στο 0. Αυτό μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμα καλό για τους καταναλωτές, αλλά σε μακροχρόνιο επίπεδο κακό για την οικονομία. Εξακολουθούν επίσης να μην γίνονται δανειοδοτήσεις προς την ε, ε, αγορά μόνο 0,3% δοθήκανε περισσότερες, ε, περισσότερα δάνεια προς επιχειρήσεις, 0,4% περισσότερο για, τις, για τα νοικοκυριά, ενώ τροφοδοτεί τις τράπεζες με 60 δισεκατομμύρια ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάθε χρόνο. Με όλα αυτά λοιπόν μπορεί να είναι θετικά για τις τράπεζες αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Λοιπόν συνεχίζεται να υπάρχει μια, ε, ένας τέτοιος συνδυασμός ο οποίος εμπλέκει τις κρατικές οικονομίες με την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χωρίς ε, διαφορετικές αλλαγές, χωρίς πραγματικές επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρξει καμία αύξηση της απασχόλησης ούτε αύξηση της οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρώπη. Κυρία Κάπελ, υπάρχει μία μπλε κάρτα του κυρίου Αρνό. Την δέχεστε, κυρία, του κυρίου συγγνώμη, δέχεστε. Ευχαριστώ. Το να εξετάσουμε αν επέτυχε ή όχι το ευρώ, το ευρώ μπορούμε να το δούμε αν συγκρίνουμε τις οικονομίες της Ευρωζώνης και τις οικονομίες που είναι έξω από την Ευρωζώνη. Οι τελευταίες έχουν αναπτυχθεί ταχύτερα από το ευρώ. Συμφωνείτε μαζί μου ότι το ευρώ είναι ένα λαθασμένο πολιτικό εγχείρημα και όχι ένα επιτυχές οικονομικό εγχείρημα. Συμφωνείτε πρέπει να δεχτούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των χωρών που δεν θέλουν να μπουν στο ευρώ και ακόμα και των χωρών που θέλουν να βγουν από το ευρώ. Συμφωνώ πράγματι ότι πρέπει να σεβαστούμε τα δημοκρατικά δικαιώματα κάθε χώρας να διαλέξει την δική της θέση. Νομίζω θα ήταν πολύ λογικό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νόμισμα, αλλά με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ενότητα για τα θέματα αυτά. Αυτό δεν υπάρχει και επομένω είναι πολύ αμφίβολα αν θα μπορέσουμε να έχουμε ένα τέτοιο επιτυχημένο νόμισμα κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Πάω να δω. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα που είχα θίξει και όταν συζητούσαμε την προηγούμενη έκθεση για την ΕΚΤ. Δηλαδή την, ε, τον δανεισμό από τράπεζες προς επιχειρήσεις. Η κατάσταση παραμένει μη ικανοποιητική σήμερα παρά τα μέτρα που έχουν αναλυφθεί τελευταίως. Οι ευρωπαϊκές ε, εταιρείες και επιχειρήσεις ε, εξαρτώνται από τον δανεισμό από τράπεζες και άλλες ε, πηγές και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Καλωσορίζω τα μέτρα της ΕΚΤ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό μεταξύ των οποίων αρνητικά επιτόκια και μακροπρόθεσμες, ε, μακροπρόθεσμες αναχρηματοδοτήσεις, στοχευμένες αναχρηματοδοτήσεις, όμως βλέπουμε από την φετινή και μόνον έκθεση ότι παράλληλες πολιτικές πρωτοβουλίε μπορεί να ήταν σχετικά αποτελεσματικές, ιδίω για τον κίνδυνο της οικονομικής σταθερότητας και να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι τράπεζες. Όμως με τις μακροπρόθεσμες ε, στοχευμένες αναχρηματοδοτήσεις και παρά τον περιορισμό των τραπεζικών δανείων τελικά δεν μπόρεσε να υπάρξει ανάπτυξη των δανείων όπως ε, είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ένα σύνολο 400 δις ε, διοχετεύτηκαν στο τραπεζικό σύστημα μεταξύ πέντε γύρων πληστηριασμών TLTO όμως ο δανεισμός από τράπεζες αυξήθηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2014 και 2015. Η έκθεση για το 2014 δείχνει ότι οι υποστατικέ συνθήκες για τι εταιρείε παρέμειναν αυστηρέ παρά ε, το γεγονό ότι σε κάποιε χώρε τη Ευρωζώνη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιε βελτιώσει. Είναι πολύ ακριβώ λοιπόν ο δανεισμό από ιδιώτε. Τα επιτόκια των τραπεζών για τον δανεισμό ε, δεν αναπτύσσουν τι πολιτικέ εξελίξει και θα πρέπει να φροντίσουμε το θέμα αυτού του δανεισμού προ τι επιχειρήσει και κυρίω τι μικρομεσαίε. Κυρία Μπερέ, ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της ε, ΕΚΤ, ξέρετε ότι η δική σας παρουσία, εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία και υπό το φως της Τρόικας ε, και της δράσης της, της Βρυξέλλες. Ε, η δράση της ΕΚΤ λοιπόν, η υλοποίηση των μνημονίων, ιδίω για την Ελλάδα, είναι κάτι που πρέπει να φωτιστεί από εσάς. Χρειαζόμαστε τις απαραίτητες αποσαφηνήσεις ασχέτως ε, της ποιότητας της νομισματικής πολιτικής που διεξάγεται, αυτή δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Χρειάζεται ανάκαμψη των επενδύσεων από καιρού εις καιρών όπως παρατηρούμε. Είπατε ο ίδιος ότι οι οικονομικές συνθήκες δεν είναι και τόσο πρόσφορες και ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση πρέπει κατεπηγόντως να ολοκληρωθεί και στο τραπεζικό της ε, σκέλος. Δεν λείπει όμως μόνο αυτό το κομμάτι, αλλά χρειάζεται και η Ένωση των ε, Κεφαλαγορών. Και πρέπει επιτέλους να περατωθεί αυτή η Οικονομική και Νομισματική Ένωση με τον συντονισμό και των προπολογισμών. Είστε ένας από τους συντάκτες της έκθεσης των πέντε προέδρων, όπου το θέμα αυτό θίγεται. Δεδομένη τη οικονομική λοιπόν κατάσταση τη Ευρωζώνη, δεδομένων των δυσχεριών εντό των οποίων βρίσκονται κάποια από τα κράτη-μέλη μα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να επιταχυνθεί λιγάκι αυτό το πρόγραμμα. Ότι η προοπτική να περιμένουμε το 2017 ώστε μαζί με την νομισματική πολιτική να οδεύει και η οικονομική πολιτική. Δεν θα πρέπει να κινητοποιηθούμε τώρα και να μην περιμένουμε τόσο πολύ. Και τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, που δεν αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Μαριά και ε, είναι το εξή. Η χρήση των φωτονομισμάτων των 500 ευρώ, ξέρετε, ότι είναι ένα θέμα που διαρκώς επανέρχεται. Ιδίω όταν μιλάμε για την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό. Διότι είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι ο δικός σας ε, οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα έπρεπε να δώσει κάποια απάντηση. Ευχαριστούμε. Κούσμιουκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, κύριε Ντομπρόφσκης, να θυμίσω κάποιες δηλώσεις του 2012 του κυρίου Ντράγκη του Ιδίου που έλεγε ότι θα κάνει whatever it takes, ό,τι χρειαστεί για να πάνε όλα καλά το ευρώ. Έκτοτε η ΕΚΤ εφαρμόζει χαμηλότατα επιτόκια, σχεδόν αρνητικά, και από το Μάρτιο του 2015 ξέρουμε ότι 60 δις ευρώ έχουν διατεθεί στην δευτερογενή αγορά. Εάν δούμε πόσο κοστίζει το χρέος όμως των περισσότερων χρεωμένων χωρών της Ευρωζώνης, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο των επιτοκίων. Πρέπει παρόλα αυτά να προσπαθήσουμε να τονώσουμε και τον κλάδο των επιχειρήσεων. Πρέπει να προλάβουμε τις ε, αγωνίες που προκαλούν οι κερδοσκοπικές επιθέσεις. Θέλουμε να γίνει κάτι λοιπόν για αυτή την απογοήτευση με την ευρωπαϊκή οικονομία που δεν αρκεί για να την τονώσει ούτε το πρόγραμμα του κυρίου Γιούνκερ για τι επενδύσει βλέπουμε ότι είναι πολύ λίγε οι καλέ επιδόσει στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή και ότι τα πάνε καλύτερα οι χώρε που δεν έχουν το ευρώ παρά αυτέ που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρά το γεγονό ότι το γενικό περιβάλλον είναι προβληματικό, οι προβλέψει για την ε, ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θετικέ, 1,7%. Παρά όλα αυτά, το υψηλό επίπεδο χρεών στα κράτη-μέλη θα πρέπει να μειωθούν περαιτέρω. Γι' αυτό χρειάζεται να υπάρξει μια καλύτερη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εξάλλου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δυνητικοί κίνδυνοι, κύριε Πρόεδρε Ντράκη, μιας πολιτικής χαμηλών επιτοκίων. Σκέφτομαι για τα θέματα των συντάξεων και των ασφαλιών. Πολλές από τις πολιτικές σας ε, παρεμβάσεις έχουν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο και εδώ καταδικάζω και τις ε, ύβρις της άκρας δεξιάς. Λόγω λοιπόν της κρίσης του χρέους, χρειαστήκατε να ακολουθήσετε μία, μη συμβατικές ενέργειες για να μπορέσετε να ενισχύσετε την νομισματική πολιτική. Μπορεί κανείς να διαφυσβητήσει την οδό που ακολουθήσετε, αλλά ο στόχος είναι σαφής και αποδεκτός από άλλους. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει τις, ε, να διαχωρίσει τις ενέργειες που έχουν να κάνουν με την νομισματική πολιτική και το εποπτικό τμήμα. Και αυτή τη στιγμή ελέγχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 122 τράπεζες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνουν με διαφάνεια. Είναι απαραίτητο λοιπόν και μέσα στον ε, νομισματικό διάλογο το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Λυπάμαι που αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ δεν το γνωρίζουν σε πολιτικό επίπεδο και οι εμπειρογνώμονες στα χρηματοοικονομικά δεν έχουν καμία πήξη στην κοινή γνώμη. Ντάλεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από ό,τι ξέρω αυτή είναι η τελευταία ετήσια έκθεση με την παρουσία του Μάριο Ντράγκη. Δεν έχει επιτύχει τους στόχους του σε επίπεδο πληθωρισμού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη από το 2013. Εδώ και μήνες ο πληθωρισμός είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Είναι προ των θυρών μας ο αποπληθωρισμός. Η ζήτηση μειώνεται, η προσφορά αυξάνει. Είμαστε ενώπιον λοιπόν μιας ε, Κατάσταση απολυθωρισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγοράζει αξιόγραφα αλλά τίποτα δεν λειτουργεί. Δεν προχωρούν τα πράγματα, αυξάνονται τα χρέη και δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, σταματήστε αυτό το πρόγραμμα, έχετε χάσει κάθε αξιοπιστία. Σας ζητώ να αντλήσετε τα απαραίτητα διδάγματα και να φύγετε. Ο Μάριο πρέπει να φύγει. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Τράκη, εφαρμόσατε τα ε, νομισματικά εργαλεία που διαθέτει η ΕΚΤΕ για την σταθερότητα σε ιδιαίτερα δύσιονες οικονομικές συνθήκες. Είναι αξιόπιστο το ευρώ και παραμένει ελκυστική η ευρωζώνη και τα τελευταία δύο χρόνια βήκανε και άλλα κράτη-μέλη στην ευρωζώνη. Για να κατοχυρωθεί ανάκαμψη στην ευρωζώνη και στην Ευρώπη χρειάζονται οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο κρατών μελών. Η υποτίμηση του, εθνικού, του νομίσματος δεν μπορεί να είναι το μοναδικό νομισματικό εργαλείο που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε τις ε, παγκόσμιες ε, προκλήσεις. Ε, κερδίζουμε χρόνο, αλλά σίγουρα δεν λύνουμε το πρόβλημα. Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να επαναπαύονται στις δάφνες τους, ακόμη και όταν πηγαίνει καλά η οικονομία. Οι οικονομίες που δεν είναι ανταγωνιστικές, που δεν μεταρρυθμίζουν, που δεν έχουν χρηστή οικονομική διαχείριση, που δεν προστατεύουν τις τράπεζες τους, δεν θα μπορέσουν να σωθούν από την, για την σταθερότητα των τιμών. Δεν αυξάνεται ο πληθωρισμός προς το παρόν και η ύφεση της οικονομίας στην Κίνα και σε άλλες αναδυόμενες αγορές ε, έχει ε, επιπτώσεις στην Ευρωζώνη που δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και με την ποσοτική χαλάρωση η ΕΚ θα πρέπει να δίνει περισσότερε πληροφορίες σε σχέση με το πώς θα εφαρμόσει το σύστημα χωρίς να επηρεάσει σημαντικά τη σταθερότητα των τιμών, του στόχου του πληθυσμού και τις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, και τέλος. Πρόεδρε Ταγκή, είπατε ότι όσοι καταρτίζουν την πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγαλύτερη πρόκληση. Δηλαδή πέρα από το ευρώ έχουμε και πιο επίγουσα κρίση την προσφυγή εκεί δίκιο έχετε, αλλά θα προσέθετα ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλες προκλήσεις και φυσικά υπάρχει προσφυγική κρίση, όμως ε, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως δικαιολογία για να σταματήσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε για την επίλυση του προβλήματος Ευρωζώνης. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν δύο μπλε κάρτες, αλλά δεν μπορώ να σα δώσω το λόγο. Περνάμε τώρα στην οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία. Υπάρχουν οκτώ οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στους οκτώ με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνατε σε ένα λεπτό. Και για να ξαναδώσουμε το λόγο σε αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη ζητήσει το λόγο, αυτό δεν έχει, το, αυτό δεν έχει νόημα. Δεν θα δώσω λοιπόν το λόγο σε αυτούς οι οποίοι έχουν σηκώσει μπλε κάρτα. Θα δώσουμε το λόγο στους οχτώ βουλευτές που ζήτησαν να παρέμβουν για ένα λεπτό ο καθένα. Ο κύριος Μαλετήτς έχει το λόγο για ένα λεπτό όμως. Ευχαριστώ. Φυσικά είναι σημαντικά και αξιόλογα τα μέτρα που παίρνετε κύριε Ντραγκή και φυσικά θέλουμε να χρησιμοποιηθούν ε, οι πόροι για τους ερευνητές ε, και για ε, να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη επιστημονικών οργανισμών. Όμως χρειαζόμαστε και μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής τόρωση του ανταγωνισμού και των επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ναι, μεν, όμως δεν επιτυγχάνεται έτσι οικονομική ανάκαμψη. Θα πρέπει λοιπόν να αυξηθούν οι επενδύσεις για τις επιχειρήσεις ε, που χρησιμοποιούν κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, κονδύλια διαθέσιμα για, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να δράσουμε εσπευσμένα για να ενισχύσουμε <clears throat> την οικονομία, την τραπεζική ένωση, την ένωση των χρηματαγορών και να ε, είμαστε δημιουργικοί. Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία. Κυρία Τόμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναβίβολα παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ε, ευρωπαϊκή οικονομία και έχει τους απαραίτητους μηχανισμούς για να εξασφαλίσει την ε, επίτευξη της οικονομικής μεγέθυνσης. Βέβαια είναι δύσκολο να έχει κανείς τα σωστά εργαλεία και να τα επιλέξει, αλλά βλέπουμε ήδη ότι όλα αυτά τα μέτρα μπορούν να αποδώσουν. Βέβαια δεν είναι απαρκή και δεν είναι αποτελεσματικά μέχρι στιγμή. Δεν έχουν αποδώσει το επίπεδο των προσδοκιών μα. Αλλά ανεξάρτητα από την επίκριση που μπορεί να έχει κανεί για τα μέτρα αυτά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν είναι επαρκή για να μπορέσουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μεταρρυθμίσει, όπω τονίστηκε και από πολλού συναδέλφου. Δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη επιτύχει στον ίδιο βαθμό στο να επιφέρουν τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε σοβαρές κρίσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μια μεγάλη ευθύνη να αποτρέψει αυτέ τι κρίσει. Καπούτο, κύριε Πρόεδρε. Όταν ξεκίνησε <clears throat> η κρίση υπήρξε μια πίεση πολιτική για νομισματική πολιτική για λιτότητα του προπολογισμού και διαρθωτικές αλλαγές. Το Σεπτέμβριο 2014 ο πρόεδρος Δράγκη ανέφερε τα μέτρα τα οποία θέλει να εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλλά η κρίση έδειξε τι δυσκολίε οικονομικέ στι οποίε βρίσκονται οι, Ευρωπα... οι Ευρωπαίοι πολίτε χωρί να διαδοθούν οι διαφορετικέ δυσκολίε. Οι συνέπειε από τι δράσει τη ΕΚΤ έχουν ε, δείξει και από τα στοιχεία τη Eurostat ότι δεν μπορεί να ε, αρκέσει η παρέμβαση στι τιμέ. Θα πρέπει ο μακροοικονομικό δημοσιονομικό συντονισμό να ε, γίνει μέσω και τη ευελιξία στο Σύμφωνο Σταθερότητα. Έτσι, ευάλωτη θέση των θεμελίων της Ευρωζώνης μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω. Με μέτρα όμως που θα είναι και κοινωνικά δίκαια. Ευχαριστώ πάντως τον κύριο Ντράγκη για την ε, προθυμία του να παρουσιάσει την οικονομική νομισματική πολιτική και να βοηθήσει στην ενίσχυση αυτής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει δύο κρίσεις παράλληλα, την κρίση του ευρώ και την κρίση των προσφύγων. Και οι δύο κρίσεις είναι, είναι δύο φαντάσματα που αντιμετωπίζει η, Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Η κυρία Μέρκελ είχε πει ότι θα πρέπει να δεχτούμε απεριόριστα ε, πρόσφυγες και να διατηρήσουμε τη ζώνη του ευρώ. Αντίστοιχα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να διατηρήσει με κάθε τρόπο τη ζώνη του ευρώ. Και στι δύο περιπτώσει απλώ κερδίζουν χρόνο. Τίποτα. Δεν αντιμετωπίζουν σε διαφορετικό επίπεδο την πραγματικότητα. Για την ε, περίπτωση των προσφύγων είναι ο πόλεμο και η ένδια που οδηγεί σε όλου αυτού του πρόσφυγε να έρχονται στι πόρτε τη Ευρώπη. Αλλά για την ε, κρίση του ευρώ τα πράγματα είναι πιο απλά. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό αντίστοιχα με τους πρόσφυγες, γιατί έχουμε μία ευρωζώνη. Η Ευρώπη είναι ο άρρωστος, ο άρρωστος ο οποίος δεν είναι στο Βόσπορο αλλά στο Αιγαίο. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να φύγει για να μπορέσει να ξαναβρει την οικονομική ανάπτυξη. Διέγας. Η ΕΚΤ εκπροσωπεί σήμερα το μεγαλύτερο κέντρο για κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τρόπο μάλιστα αδιαφανή ε, κοστίζοντας πολλά στους πληθυσμούς ξεπερνώντας τις εντολές που αρχικά του είχαν ανατεθεί. Αυτός ο οργανισμός προσθέτει την νομισματική πολιτική στην ε, εποπτεία των τραπεζών κάτι που προφανώς αποτελεί μια αντίφαση και ακόμα και στον οικονομικό συντονισμό ε, ανατρέχει στον εκβιασμό για να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν της οικονομικέ, πολιτικές, η ΕΚΤ. Τα κράτη-μέλη όμως κάνουν ότι τα εθνικά κράτη δεν μπορούν να καθορίσουν τη χρηματοδότησή τους όπω μπορούν, αλλά αναγκάζονται να δανείζονται με εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ και με τι αντάλλαγμα. Αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ απλώ σταθεροποιούν τι τράπεζε. Ε, αλλά το θεμετό ερώτημα που προκύπτει σήμερα είναι ότι δεδομένη αυτή τη συνάφεια, ποια είναι η πραγματική αποστολή τη ΕΚΤ σήμερα. Να υπάρχει ένα μακροοικονομικό πλαίσιο που να είναι σταθερό ή να εγγυηθεί την επιβίωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ευχαριστούμε. Έριξον. Ευχαριστώ. Πραγματικά τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον κύριο Τράκη, για τις προσπάθειες που κάνει η ΕΚΤΕ για να βοηθήσει ε, και να συμβάλλει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, λειτουργείται υποδειγματικά, όμως ταυτόχρονα είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τον πληθωρισμό και για την ποσοτική χαλάρωση. Τι μπορούμε να κάνουμε τελικά στο μέλλον, ποιε είναι οι δυνατότητες ε, που υπάρχουν, ούτως ώστε παραδείγματος χάρη να είναι πιο αποτελεσματικές οι δράσεις της ε, ΕΚΤ. Μπορούμε να στοχεύσουμε καλύτερα τις δράσεις ούτως ώστε τα χρήματα να διοχετευθούν καλύτερα, αποτελεσματικότερα στην πραγματική οικονομία, να λειτουργήσουν οι επενδύσεις που κάνουμε και να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΕΚΤ. Αυτό, γι' αυτό επ' θα ήθελα μια απάντηση ή δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, δύο είναι οι τρόποι που μπορούμε να λειτουργήσουμε στη ζωή με αμερόληπτα, ανεξάρτητα. Βασιζόμαστε σε δεδομένα και παίρνουμε τις αποφάσεις που είναι καλύτερες για, ε, ε, τους πολίτες. Ή αντλούμε τα δικά μας συμπεράσματα και πάση θυσία τα υπερασπιζόμαστε. Πώς μπορεί κανείς ε, να υπερασπίζεται την Ευρωζώνη. Ξέρουμε όλοι ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και ε, ε ας πάρουμε τα δεκμήρια. Ε, θα ήθελα να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Παραδείγματο χάρη, περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανάπτυξη 1,7% για το 2016, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει ανάπτυξη 2,6% και συνεχίζουμε στην έκθεση. Μιλάμε για αντιμετώπιση της ανισοβαρούς εκπροσώπησης των δύο φίλων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΕΚΤ τι πρέπει να κάνουμε. Ευτυχώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στην Ευρωζώνη και δεν θα έπρεπε φυσικά οι Βρετανοί Ευρωβουλευτέ να λένε σε άλλε χώρε τι πρέπει να κάνουν και δεν πρέπει να κάνουν. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, <clears throat> το 2012 με τον Μπασανινή, ο οποίος ήταν ε, γενικός γραμματέας στο προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας και μαζί με τον ε, ε, κύριο Ντράγκη ξεκίνησε η λογική της ποσοτικής χαλάρωσης. Ο στόχος ήταν να γίνει μια σειρά επενδύσεων στις χώρες που είχαν διαρθρωτικά ελλείμματα και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση των νέων μορφών ενέργειας ή τα σχέδια υποδομών τα οποία θα ήταν απόλυτα σίγουρα. Δεν έγινε πραγματικότητα αυτό για πολλούς λόγους. Γιατί όμως δεν θέλετε να ξεκινήσετε και πάλι μια ε, χαλάρωση, μια ποσοτική χαλάρωση στην πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντόμπ Ρόφσκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριε, κύριε Βουλευτές, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τη συζήτηση. Το Κοινοβούλιο έχει ζωτικό ρόλο να διαδραματίσει στην χάραξη των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών και ήταν πολύ θετική η αφοσίωση και η θέρμη με την οποία συζητήσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το ρόλο τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στο διάλογο με την ΕΚΤ γιατί είναι μια σημαντική συνιστόσα στη διαφάνεια και την, ε, το δημοκρατικό υπόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, ε, υπάρχει μια μακρά περίοδο πολύ χαμηλού πλωθυρισμού και πρέπει να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αυτό η ΕΚΤ σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη τη Ευρωζώνη. Είναι η στιγμή όλοι οι πολιτικοί θύνοντε να αναλάβουν ευθύνε ταυτόχρονα και να σεβαστούν την εντολή που του έχει ανατεθεί. Όμω ο αντίκτυπο αυτή τη κρίση δεν ήταν απλώ κυκλικό. Έχει και μια διευθυντική συνιστόσα και εμποδίζει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η οικονομική, δημοσιονομική και ε, νομισματική πολιτική είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Φέτος θα δοθεί προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που μπορεί να επιτρέψουν την ανάκαμψη στην, ε, ε, στον τομέα της ανάκαμψης, της οικονομικής αύξησης και της απασχόλησης. Νέες λοιπόν θέσεις με πιο περατωμένη, πιο δίκαιη εσωτερική αγορά, καθώς και μια προσπάθεια η οικονομική και νομισματική πολιτική να βαθύνει και να ενταθεί με ε, τις προτάσεις της έκθεσης των πέντε προεδριών. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντράγκη τώρα. Ευχαριστώ. κύριε, και κύριοι, ε, είμαι πολύ ευγνώμων για την σημερινή συζήτηση και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις περισσότερες ερωτήσεις ε, παρότι Λόγω χρονικών περιορισμών δεν θα μπορέσω να απαντήσω όλα τα ερωτήματα και μπορώ να σας πω ότι κάποια σχόλια και κάποια ερωτήματα ήταν ε, αμυγός ε, πολιτικής φύσης ε, και θα έπρεπε ίσως να απευθυνθείτε στους δικούς σας πολιτικούς ευθύνοντες ή και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια από τα ζητήματα. Προκύπτει από πολλά ερωτήματα που ακούσαμε πως πολλοί έχετε ενδιασμούς σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των μέτρων νομισματικής πολιτικής. Ε, θα ήθελα να προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί Επανειλημμένα είπα πως λειτουργούν αισίως ε, τα μέτρα νομισματικής ε, πολιτικής. Ε, όλοι οι δείκτες δείχνουν βελτίωση ως προς την παροχή πίστης και τις συνθήκες χρηματοδότησης. Για να σας δώσω μια πιο συγκεκριμένη ιδέα, έχουν στην Ευρωζώνη κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες πέσει τα τα ποσοστά από το 2008 μέχρι σήμερα και θα πρέπει να ξέρετε ότι συζητούμε σήμερα την έκθεση για το 2014 και έχουν έκτοτε συμβεί πάρα πολλά πράγματα πράγματα. Θα ήθελα να σας δώσω μια σαφέστερη εικόνα σε σχέση με την ε, έκθεση και την, ε, για το 2014. Μιλάμε για 8 μονάδες βάσης λοιπόν για το 2014 και από 140 μονάδες ε, και μετά που, για τις χώρες που επλήγησαν σοβαρά από την κρίση. Δεύτερον, Αυτές οι βελτιωμένες συνθήκες οδήγησαν σε υψηλότερες επενδύσεις και παροχή πίστη στην Ευρωζωνή υποστηρίζοντας λοιπόν την οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης ε, στα πλαίσια δυσμενών ε, εξελίξεων για να δώσω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το Μάιο του 2014 και πριν εξαγγελθούν τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, ε, η εξαγγελία των ε, μέτρων συνεργασίας βλέπαμε ε, για τις επιχειρήσεις ότι το ποσοστό ήταν 2,9% για τη διονελειψία ε, και ε, παρά τη συρρήκνωση μπορούμε να διαπιστώσουμε το 2015 και μετά ανάπτυξη τρίτον σταθερότητα της τιμής και ενίσχυση της αξιοπιστίας γενικότερα στην Ευρωζώνη αλλά και υποστήριξή της ευρεούσας ανάπτυξης θεωρούμε πώς. Εάν δεν είχαμε να λάβει αυτά τα μέτρα, τελικά θα είχε οδηγηθεί σε κανονικό αποπληθωρισμό ήδη από πέρυσι η Ευρωζώνη και θα είχαν μειωθεί ακόμη ταχύτερα οι τιμέ. Ε, ε, ε, έχουμε υπολογίσει, παραδείγματο χάρη, ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα μέτρα ποσοτική χαλάρωση, η ανάπτυξη θα ήταν κατά, ένα, κατά μία μονάδα χαμηλότερη σε σχέση με τη, και με τι προοπτικέ μέχρι το 2017 και το 2015 θα ήταν είναι αρνητική η ανάπτυξη, πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτά που προβλέπουμε αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα για το 2016. Ε, πολλοί ρώτησαν, μα τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, μπορώ να επαναλάβω αυτά που είπα και στη συνέντευξη τύπου. Με την ε, υιοθέτηση αυτών των μέτρων και τη χορήγηση χρημάτων στην πραγματική οικονομία, δεν ήταν θεαματικά τα αποτελέσματα, αλλά ήταν πραγματικά. Και τον Ιούνιο του 2014 με το πακέτο μέτρων ευνοήθηκαν ιδιαίτερω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει διότι τα ποσοστά δανειοληψία για τι μικρέ επιστώσει μειώθηκαν περισσότερο από ότι για τα μεγάλα δάνεια. Και ξέρετε, υπάρχουν δύο είδη υπηρεσιών, δηλαδή η δανειοδοσία των τραπεζών. Ρωτάμε εμεί τι Τράπεζε, τι σκοπεύετε να κάνετε, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντε που θα συνυπολογίσετε για να αποφασίσετε αν θα χορηγήσετε ένα δάνειο ναι ή όχι. Η απάντηση είναι ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει τέτοιος ε, παράγοντας ε, περιορισμού ε, της δανειοδοσίας αυτή τη στιγμή και υπάρχει και μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και βάσει της οποίας βλέπουμε για την πρόσβαση των ΜΜΕ στη δανειοδοσία ε, ότι υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία από πλευρά των τραπεζών για το εξάμεινο από μέχρι το Σεπτέμβρη το 2015. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία βεβαίως τα ποσοστά δανεισμού για τα ιδιαίτερα μικρά δάνεια είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τα ε, μεσαία δάνεια, κυρίω σε φαθέστερε οικονομίε τη Ευρωζώνη. Και φυσικά αυτό δείχνει και το μεγαλύτερο κίνδυνο ε, τη ε, δανειοδοσία προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Έχουμε επίγνωση του κινδύνου συγγνώμη, και θα προσπαθήσουμε να τον υπερβούμε. Και φυσικά δεν έχουμε επιτύχει ε, όλα τα ευθεία και φυσικά πρέπει να κάνουμε περισσότερα και φυσικά θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω οι συνθήκες ε, ε, δανειοληψίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως προς την νομισματική μας πολιτική, όπως σας είπα και στην εισαγωγική μου παρουσίαση, επειδή υπάρχει και ελοχεύει ακόμα αυτός ο κίνδυνος σε σχέση με τη σταθερότητα των τιμολόγων της ύφεσης οικονομίας, ε, βάσει της εντολής της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται ενδεχομένως να αναθεωρήσει στις αρχές Μαρτίου την νομισματική της πολιτική ανάλογα και με τα στοιχεία που θα λάβουμε και τις προβλέψεις διάφορα ερωτήματα, διάφορες δηλώσεις που έγιναν σχετίζονται με τους πιθανούς κινδύνους των χαμηλών επιτοκίων και των ε, μη αντισυμβατικών μέτρων που έχουμε αναλάβει, κυρίως σε σχέση με την θεωρία ότι τα χαμηλά επιτόκια πλήττουν ε, τους ε, αποταμιευτές και ότι η πολιτική μας μπορεί να απειλήσει την σταθερότητα των τιμών κυρίως τα συνταξιδοτικά ταμεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες και γενικότερα τους ε, αποταμιευτές. Ε, το έχουμε συζητήσει αυτό επανειλημμένα. Θα ήθελα όμως να τονίσω το εξή. Για τις αποταμιεύσεις, αληθεύει ότι τα ονομαστικά επιτόκια για τις ε, αποταμιεύσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλά, ιστορικά χαμηλά. Επίσης, εξηγήσω ότι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων αντικατοπτρίζει τις οικονομικές και διαρθρωτικές συνθήκες της εποχής. Και αν με ρωτήσει κανείς πόσο θα κρατήσει, η απάντηση είναι θα κρατήσει μέχρι ότου βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον. Άρα η χαμηλή απόδοση των αποταμιεύσεων είναι όχι αιτία, αλλά ε, αποτέλεσμα αιτιατό του δεδομένου αυτού. Χαμηλό δυναμικό και ε, σόρευση πόρων. Αν Φερρυπίν απίσχαμε από την ε, κοινοτική αυτή επιλογή. Τι θα γινόταν. Ναι, δύσκολο να φανταστεί κανεί ότι θα περικόπταμε ακόμη περισσότερο τον οικονομικό δυναμισμό και εν τέλει θα συμβάλαμε στην παράταση μιας περίοδου χαμηλών επιτοκίων με περαιτέρω ύφεση. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει και να σημειώσουμε ότι οι καταθέσεις δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ε, ο πολίτης προστατεύει την αποταμιευσή του. Αν κοιτάξουμε τα δεδομένα των οικοκυριών, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα οικονομικά στοιχεία τα οποία μπορούν να προστατεύσουν την αποταμίευση. Μια πρόσφατη μελέτη της Bundesbank δείχνει πραγματική απόδοση σε χαρακτηριστικό χαρτοφυλάκιο οικιακό από το 2008 με αύξηση 1,5% χαμηλότερη βεβαίως από το μέσο όρο προ-κρίσεως... αλλά ασφαλώς πολύ ψηλότερο από άλλες περιόδους, περίπου της δεκαετίας του 90. Άρα δεν μπορούμε να μιλούμε για απαλωτρίωση καταθέσεων, όπως έχουν πει κάποιοι σε άλλες περιστάσεις, όχι σήμερα. Εν τέλει, πιθανές συνέπειες για τον καταθέτη. Ε, αυτές πρέπει να τις κοιτάξουμε σε ευρύτερο πλαίσιο οι καταθέσεις προκύπτουν από εισόδημα που πρέπει να κερδίσει ο πολίτης με την υποστήριξη και της απασχόλησης και των επενδύσεων μέσα σε συνθήκες κατάλληλες. Η νομισματική μας πολιτική ως εκ τούτου υποστηρίζει τη δυνατότητα να αποταμιεύει κανείς. Επίσης, ανησυχίες εκφράστηκαν για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τον τρόπο με τον οποίο η νομισματική μας πολιτική μπορεί να την επηρεάσει. Η σταθερότητα των τιμών είναι προϋπόθεση, βάση για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και πρέπει να εμείνουμε σε αυτό το στόχο ταυτόχρονα οι, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής μπορεί να έχουν ε, μη προσδοκόμενα παρεμπίπτοντα σε συνέπειες. Για να τις αντιμετωπίσουμε όμως χρειάζονται και μακρο και μικρο οικονομικά μέτρα ως εργαλεία, όχι αλλαγές στην νομισματική πολιτική. Και σύντομα θα ήθελα τώρα ένα σχόλιο να διατυπώσω για την εμπλοκή της ΕΚΤ στα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής εν γέννη, ένα άλλο από τα σημεία που επισημάνθηκαν. Όταν σχηματίστηκε η Τρόικα στις αρχές του 2010, δεν είχε εξοπλιστεί ακόμη η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση με την δυνατότητα αντιμετώπισης της απώλειας πρόσβασης αγορές για τα κράτη και Αρχικά είχε σχεδιαστεί ο συμβουλευτικό ρόλο τη ΕΚΤ, όπω και τη Επιτροπή και του Δονοτού από τα κράτη και για την Ελλάδα. Και είχε θεωρηθεί ότι συμπληρώνει χρήσιμα η παρουσία μα ε, ένα πρόγραμμα στεναρό. Δηλαδή η Τρόικα θα προσέφερε την εμπειρία των θεσμών στα κράτη ως υποστήριξη. Και υπήρχαν ε, σαφείς λόγια τους οποίους ζητήθηκε η συμβολή της ΕΚΤ προκειμένου να λειτουργήσει το πρόγραμμα, αλλά και γιατί απεδέχθη η ΕΚΤ. Γιατί αυτό θα σημαίνει έναν η επιτυχία των προγραμμάτων θα σημαίνει έναν καλό μηχανισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ο σχεδιασμός αυτός κωδικοποιήθηκε, σημειώνω και υπογραμμίζω, με την συμφωνία ESM και με το TUPAC από τους συνομοθέτες του ΔΕ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επικύρωσε την νομιμότητά της. Ως εκ τούτου η ΕΚΤ προσφέρει μέσα μέσω των προγραμμάτων της Συμβουλές της σε πέντε κράτη-μέλη έκτοτε. Δεν πρέπει ωστόσο να λησμονούμε ότι η τελική επιλογή, οι αποφάσεις, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων ανήκει στο Eurogroup, τους Υπουργούς των Οικονομικών και τον Μηχανισμό ESM, όχι στους θεσμούς που εμπλέκονται στο πρόγραμμα. Και όπως είπα και σε άλλες περιστάσεις, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα είναι ίσως για πάντα μέρος της Τρόικα. Ωστόσο, πρέπει πολύ προσεκτικά να σχεδιαστεί η κατάλληλη χρονική στιγμή για την αλλαγή της σύνθεσης και αυτό δεν είναι δική μου, δικό μου καθήκον. Μερικές παρατηρήσεις τώρα σε σχέση με τη διαφάνεια. Και σημειώνω εδώ ότι το 2015 ήταν έτος με πληθώρα αποφάσεων που είχαν ως στόχο τη βελτίωση της διαφανείας μας και ασφαλώς τα όσα κάναμε ενισχύουν και την προσήλωσή μας. Η δημοσίευση των απολογισμών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το υποπτικό Συμβούλιο όπως και εγώ δημοσιεύουμε αυτά τα στοιχεία σε ένα στόχο βελτίωσης της διαφάνειας. Ταυτόχρονα είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε περαιτέρω πληροφορίες σε ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, υπογραμμίζοντας έτσι ότι είναι διαφανές όργανο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από το Σεπτέμβριο του 2015, παραδείγματι, οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες μπορούν να κοινοποιούν ζητήματα σχετικά με τον ELA στις τράπεζες των χωρών τους, όπου θεωρούν ότι μια τέτοια κοινοποίηση είναι απαραίτητη προσφέρουμε και εμείς επιπλέον πληροφορίες για το σχεδιασμό μας. Τα σχέδια παραδείγματι για την συλλογή των anacredits, των στοιχείων δηλαδή για μακροπρόθεσμο δανεισμό. Και έτσι οι εξελίξεις και στη διαχείριση και στην πρόσβαση στα έγγραφα ενισχύει και τη διαφάνεια και τη διάθεση για λογοδοσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύντομα για την ολοκλήρωση της, της Νομισματικής Ένωσης τώρα. Όπως θα έχετε σημειώσει, η έκθεση των πέντε προέδρων αποτελεί έναν οδικό χάρτη για την πρόοδο προς περισσότερη ολοκλήρωση και βεβαίως είναι ευπρόσδεκτη και η πρόσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βραχυπρόθεσμα μέτρα που πρέπει πλέον να υλοποιηθούν πλήρως. Για την έκτη ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης βεβαίως έχει ε, ε, υπέρτατη σημασία και αυτό σημαίνει ότι κοινοί κανόνες, κοινά συμφωνημένοι κανόνες θα πρέπει και να εφαρμόζονται. Κύριο παράδειγμα του που θα πρέπει ιδιαίτερα να δοθεί έμφαση για πρόοδο είναι η υλοποίηση της BRRD και της TGST σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ακόμα δεν υπάρχει κοινό σημείο για το, ε, για το κοινωνικό ταμείο, κοινό ταμείο ε, εκαθαρίσεων. Επίσης, δεν έχουμε κοινά στοιχεία, κοινές λύσεις για ένα σχέδιο κοινού ταμείου εγγύησεων των καταθέσεων. Αυτό γιατί, γιατί υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις από τα κράτη και στην Τραπεζική Ένωση και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να ε, λυθούν πολλά προβλήματα της νομισματικής μας ένωσης. Για να εφαρμοστούν όμως οι βραχυπρόθεσμες προτάσεις της εκθέσεως των πέντε προέδρων, ε, που είναι βέβαια μια απαραίτητη συνθήκη αλλά όχι επαρκή τη Ένωση, θα πρέπει να κρατεθούν και οι προτάσεις για τα μακροπρόθεσμα ζητήματα. Και θα ήθελα, όπως έχω και άλλες φορές πει, να υπογραμμίσω ότι για την ευημερία της Ευρωζώνης, και εδώ θα συμφωνήσω με κάποιες τις παρατηρήσεις σήμερα, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στην νομισματική πολιτική. Η νομισματική πολιτική δίνει τον απαραίτητο χώρο. Είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής όπως είπα συνθήκη για την ανάκαμψη. Ώστε να γίνει η ανάκαμψη δηλαδή διαρθρωτική σε σχέση με αυτό που είναι τώρα που είναι απλώς κυκλική. Μια ερώτηση σχετικά με τα χαρτονομίσματα, τα μεγάλα χαρτονομίσματα για τα μεγάλα ποσά. Και θέλω να πω ότι το εκτελεστικό μας συμβούλιο έχει εξετάσει το θέμα αυτό πολλές φορές και εξετάσει και τεχνικά το ζήτημα των μεγάλων χαρτονομισμάτων. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε απόφαση. Υπάρχουν ζητήματα για το πώ μπορεί να υλοποιηθεί, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να υλοποιηθεί μια τέτοια απόφαση, αλλά και πώς θα πρέπει να κοινοποιηθεί, ποια θα είναι η επικοινωνιακή επιλογή. Θέλουμε τις αλλαγές να τις κάνουμε με τρόπο τακτό και σας διαβεβαιώ ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε έναν χώρο άνεσης για τους εγκληματίες. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντράγκη. Ο εισηγητής για δύο μόλις λεπτά, ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους <clears throat> για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση. Κύριε Ντράγκη, συμφωνώ ότι πρέπει να δούμε το μέλλον αυτό όμως προϋποθέτει ότι πρέπει η του να δει τα λάθη της στο παρελθόν. η ΕΚΤ υποτίμησε τους κινδύνους αποπληθωρισμού και μόνο το σεπτέμβριο του 2014 ξύπνησε και κατέφυγε σε μη συμβατικά μέσα σχεδιάζοντας ποσοτική χαλάρωση την οποία τελικά άρχισε να εφαρμόζει από τον ιανουάριο του. 2015. χιλιάδες επίσης αργήσατε να μειώσετε τα επιτόκια όπως έκανε έγκαιρα η fed και δεν απαντήσατε κύριε ντράγκη γιατί ακόμη η ανεργία βρίσκεται στα ύψη ταυτόχρονα συνεχίσατε να επιμένετε στη σκληρή δημοσιονομική πολιτική και στη λιτότητα. δεν απαντήσατε κύριε ντράγκη για τα μέτρα που πρέπει να λάβετε για να σταματήσει η σύγκρουση συμφερόντων εντός της ΕΚΤ. τελικά πότε θα φύγετε από την τρόικα κύριε ντράγκη όπως σας υπέδειξε το δικαστήριο της ευρωπαϊκής ένωσης στην απόφαση σε 62 του 2014 και εμέσως πριν λίγο κι εσείς ο ίδιος το δεχτήκατε. τελικά πώς εξηγείτε κύριε ντράγκη οι δανειζόμενοι ελλάς να δανείζει μέσω από την ποσοτική χαλάρωση με την τράπεζα της ελλάδος 17 δισεκατομμύρια ευρώ στους δανειστές της. Πού βρήκε ο κύριος Τουρνάρας 17 δισεκατομμύρια ευρώ και συμμετείχε η Τράπεζα της Ελλάδος στην ποσοτική χαλάρωση το 2015 δεν απαντήσατε κύριε ντράγκη για τον τρόπο εφαρμογής των μνημονίων. νύπτετε τα σχήρα σας ως πόντιος πιλάτος ρίχνετε τις ευθύνες στο eurogroup όμως εσείς προσπαθήσατε και επιβάλατε πιστωτική ασφυξία στην ελλάδα το 2015 και επιβλήθησαν τα capital controls. η εκβιαστική σας πολιτική και η στήριξη των δανειστών προκειμένου να καμφθεί το όχι του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα του ιουλίου του 2015 καταγράφεται ως μελανό σημείο της ΕΚΤ ως απαράδεκτη παραβίαση της λαϊκής κυριαρχίας στην ελλάδα ως κατάλυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. κύριε ντράγκη για να υπάρξει πράγματι η λύση των αντιφάσεων στην ευρωζώνη πρέπει η ευρωζώνη να πάψει να είναι ένωση δανειστών. πρέπει να επιληθεί το θέμα του δημοσίου χρέους και αυτό πρέπει να γίνει με διαγραφή του επονίδη του χρέου και αμοιβαιοποίηση του χρέου. τα παραπάνω σημεία υπήρχαν στην αρχική εισήγηση αλλά το epp και το sd και το alde φρόντισαν να αφαιρέσουν την κριτική προς την ΕΚΤ. όπως είπα ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως δηλαδή ήταν πιο ντραγκιστές και από εσάς κύριε ντράγκη. ευχαριστώ.